Συνάδελφοι και συναδελφέ, σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με την Κυπρία Υπουργό Εξωτερικών. Με μεγάλη χαρά την καλωσορίζω, την κυρία Κοζάκο Μαρκουλή. Και περιμένουμε μεγάλη επιτυχία από την Κυπριακή Προεδρία. Έχουμε πολλά σοβαρά θέματα που πρέπει να λυθούν και ελπίζουμε να λυθούν από την Προεδρία αυτή. Πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ένωσης, ιδιαίτερα για τα χρηματοπιστωτικά, αλλά θα θέλαμε ως Επιτροπή Εξωτερικών να τονίσουμε και τη σημασία της διαδικασίας της διεύρυνσης που θέλουμε να συνεχιστεί Ξέρουμε ότι είναι και δική σας προτεραιότητα, της Προεδρίας σας δηλαδή. Θα σας δώσω τώρα την ευκαιρία να μας πληροφορήσετε για τις προτεραιότητες σας γενικότερα και μετά θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Thank you, Mr. Uh, Chairman. Uh, uh, Στην αρχική μου παρουσίαση θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα κατά τη διάρκεια των uh, ερωτοαπαντήσεων και της ανταλλαγής απόψεων θα χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα. Ε, πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ιδιαίτερη η τιμή να βρίσκουμε σήμερα εδώ μαζί σας με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία για να παρουσιάσω ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτή συγκεκριμένα τις προτεραιότητές μας κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Θέλω να τονίσω από την αρχή το σημαντικό ρόλο που προσδίδουμε ως Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ισότιμο συνομοθέτη. Στόχος μας είναι η συνεχής επαφή και συνεργασία μαζί σας με γνώμονα την προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Βασικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας είναι η προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη, η οποία πρέπει να εξέλθει ενισχυμένη από την τρέχουσα οικονομική κρίση και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Η διεύρυνση αποτελεί μία από τις κυριότερες μας προτεραιότητες, αφού συμβάλλει έμπραχτα και προς το στόχο για μια καλύτερη Ευρώπη, ως μια διαδικασία που αναδεικνύει αφενός τις οικουμενικές αξίες του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και αφετέρου την ίδια την Ένωση ως καταλήτη στην εμπέδωση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της σταθερότητας και της ευημερία σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου στοχεύουμε την επίτευξη απτής προόδου σε όλες τις επιμέρους συναφείς πτυχές της πολιτικής της διεύρυνσης. Καθοδηγητικές μας γραμμές θα είναι οι αρχές της αυστηρής αιρεσιμότητας και ότι η κάθε υποψήφια κρίνεται σύμφωνα με την αξία της. Απαρέγκλητη μας θέση είναι ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καμία περίπτωση δεν σταματά με την ένταξη της Κροατίας την 1η Ιουλίου 2013 και ότι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί με την ευκαιρία αυτή την προσχώρηση κράτους για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια θα πρέπει να τύχει της δέουσας εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς βέβαια και της Ισλανδίας και της Τουρκίας, θα είναι μίζωνος σημασίας για την Προεδρία μας. Όσον αφορά την Κροατία, κοινή αντίληψη είναι ότι οι προετοιμασίες της για ένταξη βαίνουν ομαλώς. Προτιθέμεθα να παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες της Κροατίας για εκπλήρωση των συστάσεων της Επιτροπής εν ώψη και της υποβολής από την Επιτροπή της συνολικής έκθεσης παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το φθινόπωρο. Αναφορικά με το Μαυροβούνιο, χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και τονίζω την απόλυτη ετοιμότητα και αποφασιστικότητά μας για επίτευξη ουσιώδους πρόοδου επί αυτών. Εξίσου σημαντική αξιολογούμε παράλληλα την απόφαση για απόδοση καθεστώτος υποψήφιου προσένταξη στη Σερβία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 1η Μαρτίου 2012. Η πράξη μας αυτή αναμφισβήτητα αντανακλά την πρόοδο που επιτελέστηκε από την Σερβία στον τομέα των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων καθώς και την πλήρη συνεργασία της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Υπογραμμίζω την πρόθεσή μας για προσεκτικό χειρισμό της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας, προσβλέποντας ότι θα αναφύουν οι απαραίτητες συνθήκες για λήψη απόφασης έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, εφόσον βεβαίως προϋπάρξει θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσεβόδοση αυτών των προσπαθειών είναι κρίσιμη σημασίας όπως η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί στη Σερβία θα παραμείνει σταθερά προσιλωμένη στο στόχο της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της χώρας. Σε σχέση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως Προεδρία προσβλέπουμε ότι οι κατάλληλες εξελίξεις στο ονοματολογικό θα επιτρέψουν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη χώρα, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ως θέση του Συμβουλίου την σημασία διατήρησης καλών σχέσεων γειτονίας. Αναφορικά με την Αλβανία, κοινή αντίληψη είναι ότι επιβάλλεται η εκπλήρωση των 12 κεντρικών προτεραιοτήτων ως προς την περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Όσον αφορά την Βοσνία Ερζεγοβίνη, η διαδικασία μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να συνεχιστεί καθώς και να υπάρξει συμμόρφωση για την απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Φίντσι. Πρόοδος σε αυτό το ζήτημα θα λειτουργήσει καταλητικά ως προς την υποβολή μιας αξιόπιστης αίτησης για ένταξη της χώρας, ελπίζουμε, κατά την διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Παρά την σταθερή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μία αναγνώριση της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας από το Κωσυφοπαίδιο, επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την περίοδο της Προεδρίας της θα ενεργεί με αντικειμενικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη πλήρως και ισότιμα τις θέσεις όλων των εταίρων της. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα καταβάλουμε εξάλλου κάθε προσπάθεια για να δοθεί η ισχυρότερη δυνατή όθηση στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, η οποία αδιαμφισβήτητα προχωρεί με σταθερούς ρυθμούς από την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεών της. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των εναπομεινάντων προς άνοιγμα κεφαλαίων του κεκτημένου συγκαταλέγονται θέματα ιδιαίτερης ευαισθησίας, τα οποία επιβάλλουν λεπτούς χειρισμούς προτιθέμεθα να ενεργήσουμε ως έντιμοι μεσολαβητές με μοναδικό στόχο την εξέβρεση αμοιβαίως αποδεκτών φόρμουλων πάντοτε στα πλαίσια της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Σε σχέση με την Τουρκία, παρά τη γνωστή σε όλους προκλητικότατη και προσβλητική συμπεριφορά της έναντι ενός θεσμού του θεσμού της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόθεσή μας παραμένει η παρακολούθηση και προώθηση της πορείας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Η προσέγγιση μας θα είναι αντικειμενική και πραγματιστική και θα εδράζεται στις καθιερωμένες πρακτικές και διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για όλες τις υποψήφιες χώρες. Ταυτόχρονα θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της θετικής ατζέντα ως προνοείται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή ότι η εν λόγω διαδικασία είναι υποστηρικτική της διαπραγματευτικής διαδικασίας σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα οικεία συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει εξάλλου μεγάλη σημασία και προτίθεται να ενεργήσει αναλόγως στην προώθηση της επεξεργασίας του νέου κανονισμού για το μέσο προεταξιακης βοήθειας στοχεύοντας την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός αυτού του εξαμήνου. Επιπρόσθετα, το φθινόπωρο του 2012 η Κυπριακή Προεδρία θα έχει την ευθύνη της συζήτησης στο Συμβούλιο επί του πακέτου διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012. Όπως κάθε Προεδρία θα εργαστούμε με συνέπεια για υιοθέτηση ισορροπημένων και αντικειμενικών συμπερασμάτων, τα οποία θα αντανακλούν πιστά τις θέσεις όλων των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα υποβοηθήσει, όποτε καταστεί αναγκαίο, στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της υπάτης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπως και της εξωτερικής υπηρεσίας ευρωπαϊκής δράσης. Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Προεδρία θα στηρίξει τις προσπάθειες της υπάτης εκπροσώπου αναφορικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και ιδίως την νότια διάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίξει την εκδημοκρατικοποίηση των νότιων εταίρων μας. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθεί ο εμπορικός και οικονομικός διάλογος με τις χώρες της περιοχής καθώς και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η μετανάστευση, η κινητικότητα και η ασφάλεια. Ταυτόχρονα η Κυπριακή Προεδρία θα συμβάλλει στις προσπάθειες της υπάτης εκπροσώπου για την προώθηση των στόχων εξίσου σημαντικής ανατολικής εταιρικής σχέσης. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ο στόχος θα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα εντός του πλαισίου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 2020, που θα επιτρέψει επίσης τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γειτονικές χώρες και άλλους εταίρους. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτό το θέμα θα είναι συνεχής. Η Κυπριακή Προεδρία θα στηρίξει επίσης τις προσπάθειες της υπάτης εκπροσώπου για την εδραίωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στρατηγικούς εταίρους μας και για την προώθηση των σχέσεων της Ένωσης με ανερχόμενους παγκόσμιους παράγοντες. Θα ήθελα να σταθώ για λίγο στις ραγδαίες εξελίξεις στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Η Κύπρος ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας άριστες σχέσεις με όλους τους Άραβες γείτονές της αλλά και με το Ισραήλ μπορεί να συμβάλλει μέσα και από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των ευρωπαϊκών θέσεων στην περιοχή. Οι αλλαγές στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης είναι κοσμογονικές. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της με γνώμονα τη σταθερότητα και τον εκδημοκρατισμό της περιοχής σεβόμενοι πάντοτε τις εσωτερικές διαδικασίες των χωρών αυτών. Οι εξελίξεις στον αραβικό κόσμο επηρεάζουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης, οικονομίας και άλλα. Γι' αυτό και σε συνεννόηση πάντοτε με την υπάτη εκπρόσωπο θα συμβάλλουμε στη συνέχιση του οικοδομητικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Καταληκτικά, θα ήθελα να τονίσω εκ νέου την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στον ανδιαφυσβήτητα ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η επιτυχής διεκπεραίωση των προαναφερθέντων στόχων και προτεραιοτήτων θα εξαρτηθεί και από το επίπεδο της στενής συνεργασίας μας με τον ίδιο τον θεσμό του Κοινοβουλίου, των Επιτροπών, των Υπηρεσιών και βεβαίως των μελών του. Να είσαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσουμε προς, την, προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την προσωπική σας δέσμευση και την δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας για να προωθήσει τους στόχους της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα της ε, διεύνησης και της πολιτικής γειτονίας προς τα νότια και προς τα ανατολικά. Θα ήθελα τώρα να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους μου να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ξεκινώ με τον κύριο Σαλαφράγκα. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καλώ ήλθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία σας εξ ονόματο του ΕΛΚ. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Εγώ ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση από τα εισαγωγικά σας λόγια, ιδίως σε ό,τι αφορά το λόγο, τον ρόλο μάλλον που αποδίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν συννομοθέτη. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να αντιμετωπίσετε όλες τις διεκδικήσεις του Κοινοβουλίου ή να ε, κατά κάποιο τρόπο να κολακεύσει τη ματαιοδοξία του, αλλά σίγουρα το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε διεθνές επίπεδο, προβλήματα τα οποία μας εγκαλούν όλους και ελπίζουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Υπουργέ, εγώ έχω καταγράψει αυτά που αναφέρατε, τον, την καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου και της ΥΠΑ του εκπροσώπου, ακολουθώντας την πραγματιστική αυτή κατεύθυνση που αναφέρατε για τις σχέσεις με την Τουρκία, θα ήθελα να ξέρω αν έχετε σαν στόχο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσετε στις διαπραγματεύσεις γνωρίζοντας φυσικά ότι αυτό θα απαιτήσει και μια θετική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Αυτά που είπατε για το Μαυροβούνιο επίσης έχουν θετικό αντίκτυπο σε εμά. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα της Μακεδονίας, λέει ο Η Μακεδονία είναι μια χώρα που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με την Κύπρο. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο είναι πρόθεσή σα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα να προχωρήσετε σε μια επισημοποίηση των σχέσεων, παρά το γεγονό ότι υπάρχει φυσικά το θέμα του ονόματος και υπάρχουν και θέματα τιμερή που εμπλέκουν τη χώρα αυτή. Εάν λοιπόν μπορείτε να βρείτε μια φόρμουλα ώστε να προχωρήσετε στι σχέσει Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή. Τέλος, κυρία Υπουργέ, ε, γνωρίζουμε τις προσπάθειες της ΥΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία για τα νότια και τα ανατολικά. Θα ήθελα να γνωρίσω ποια είναι η θέση σας σε σχέση με το πρόβλημα της Συρίας, το οποίο τόσο μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας την Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και να ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία για την οποία ξέρω ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και προετοιμασία από την Κύπρο, οπότε νομίζω υπάρχουν οι καλύτερες προοπτικές για ένα πολύ πετυχημένο εξάμεινο. Κυρία Υπουργέ, αναφερθήκατε στις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Προεδρία και είναι γεγονός ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα θέματα ε, και στην περιοχή μας αλλά και διεθνώς. Αναφερθήκατε διεξοδικά στο θέμα της διεύρυνσης ε, σαν μία από τις προτεραιότητες, το οποίο έτσι και αλλιώς η Επιτροπή αυτή είναι απόλυτα σύμφωνη, γιατί είναι και από τις δικές μας τις μεγάλες προτεραιότητες. Θα ήθελα να ε, ζητήσω λίγο περισσότερο την γνώμη σας στα θέματα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στο θέμα της Συρίας. Αναφερθήκατε στην πολιτική της νότιας γειτονίας, με όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχει, στο Παλαιστινιακό, ε, ε, στα άλλα προβλήματα της περιοχής, αλλά νομίζω αυτό στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να απαντήσει με επιτακτικό τρόπο είναι η συνεχιζόμενη σφαγή στη Συρία και η τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί εκεί. Τα γεγονότα με την κατάρριψη του τουρκικού αεροπλάνου πριν καμιά-δύο εβδομάδες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Και η Προεδρία σας, παρά τις καλές σχέσεις που έχει με όλες τις χώρες περιοχής, έχει ένα μεγάλο βάρος στο να μπορέσει να είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά, ένας έντιμος συνομιλητής με στις χώρες περιοχής. Θα ήθελα λίγο την εκτίμησή σας για τα γεγονότα της Συρίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόπα. Ακολουθώντας τη σειρά των πολιτικών ομάδων δίνω το λόγο στον κύριο Μάιερ, μην ακολουθώντας μάλλον τη σειρά των πολιτικών ομάδων. Κύριε Μάιερ. Καλώ ήλθατε κυρία Μαρκουλή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να σας ευχηθώ και στην Κυπριακή Κυβέρνηση που ασκεί την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε επιτυχία. Οι θέσεις που παρουσιάσατε σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα την πολιτική διεύρυνση μου φάνηκαν πολύ ορθές και γνωρίζω ότι η Ισπανική κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα της μη αναγνώρισης του κοσυφοπεδίου έχει την ίδια ε, βάση μαζί σας. Ξέρουμε ότι μια τέτοια αναγνώριση θα σήμαινε για μας μια αναγνώριση του διεθνούς δικαίου και θεωρούμε ότι πρέπει το διεθνές δίκαιο να διέπει τις ε, διεθνείς σχέσεις και η χάρτα των ε, Ηνωμένων Εθνών να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στάση. Επίσης, νομίζω ότι η σόφρον στάση σας και η πραγματιστική σας στάση έναντι των προκλήσεων της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της ε, Κυπριακής Προεδρίας δεν θα πρέπει να μας κάνει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία θα πρέπει να γίνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον όρο φυσικά ότι θα εκπληρώσει τα απαιτούμενα για κάτι τέτοιο. Και εξάλλου δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει ακόμα το βόρειο τμήμα της ε, Κύπρου και συνεχίζει μια πολιτική επικισμού στο βόρειο τμήμα της Κύπρου που είναι απόλυτα απαράδεκτη από την άποψη του διεθνούς δικαίου. Και είναι σαφής η θέση της πολιτικής μου ομάδας στα θέματα αυτά. Ζητούμε πάντα ότι η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει τη στρατιωτική κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού και την πολιτική επικισμού ώστε να υπάρξουν οι δυνατότητες να μπορέσει να ξεπεραστεί αυτή η διαμάχη και η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. Όπως και οι συνάδελφοί μου θα ήθελα να γνωρίσω όχι μόνο για τη Συρία αλλά και επίσης και για την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας, τι αντιμετώπιση θα έχετε για την Παλαιστίνη. Και επίσης ήμουνα με τον Φερνάντο Λούγο, με τον νόμιμο πρόεδρο τη Παραγουάης την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι απόλυτα απαράδεκτη που έλαβε χώρα στην Παραγουάη γιατί ο πρόεδρος εκλέγεται από τον ίδιο το λαό της χώρας του. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω μέσα στα πλαίσια αυτά ποια θα είναι η στάση της Κυπριακής Προεδρίας αν θεωρείτε ότι είναι νόμιμες και θεμητές οι διαμαρτυρίες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό ε, στην Παραγουάη και κατά πόσο θεωρείτε ότι πράγματι η Λατινική Αμερική αποτελεί ένα στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον κύριο Μάιερ που τον προσκαλώ να με αντικαταστήσει, αλλά θα δώσω προηγουμένως το λόγο στον κύριο Βάτσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να καλωσορίσω την κυρία Υπουργό εδώ και να της ε, θέσω κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, κυρία Υπουργέ, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η άποψή μου είναι ότι και δεν είναι η άποψη τη πολιτική μου ομάδα κατά ανάγκη, ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την Κυπριακή Προεδρία. Αναρωτιέμαι κατά πόσο θα μπορούσατε να διερευνήσετε συγκεκριμένου τομεί όπου θα μπορούσε να εμφανιστεί μια καλή θέληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Άγκυρα και να του παροτρύνει να έχουν μια τέτοια επικοδομητική στάση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι η συνεχιζόμενη διαίρεση τη Κύπρου υποσκάπτει την ε, ευρωπαϊκή και διεθνή αξιοπιστία της Κυπριακής Προεδρίας και πώς μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα αυτό. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο θεωρείτε ότι, άλλα ότι τα άλλα κράτη-μέλη κατανοούν πλήρως και αξιολογούν θετικά την ειδική σχέση της χώρας σας με τη Μόσχα. Και τρίτον θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε και κατά πόσο έχετε σαν στόχο να διαπραγματευτείτε και να υπογράψετε μια εταιρική σχέση για την ειρήνη μαζί με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριε Βουάτσον. Η κυρία Λούνατσοκ έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων να σας καλωσορίσω Υπουργέ. Η επιθυμία σας να έλθετε σε επαφή μαζί μας και ελπίζω να επαναληφθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Θα αναφερθώ σε θέματα στα οποία ήδη αναφέρθηκαν άλλοι συνάδελφοι μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βουάτσον για την ειδική σχέση της Κύπρου με τη Ρωσία, ιδιαίτερα σχετικά με την κατάσταση σήμερα στη Συρία. Πιστεύετε εσείς ότι λόγω αυτής της ειδική σχέσης που έχετε με τη Ρωσία να μπορέσετε να παίξετε έναν κάποιο ρόλο ενδιαμέσου θα έλεγα σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς στη Συρία, ο Ασάντ δολοφονεί τους πολίτες του, Ξέρουμε τις προσπάθειες που γίνονται και από τα Ηνωμένα Έθνη και να παρατηρήσω εδώ ότι πριν μερικούς μήνες ένα ρωσικό πλοίο με όπλα πήγαινε στον Ασάντ μέσω της Κύπρου και από ό,τι κατάλαβα οι κυπριακές αρχές δεν του το απαγόρευσαν παρότι υπάρχει απαγόρευση πωλήσεως όπλων από τα Ηνωμένα Έθνη εις βάρος του Ασάντ. Γιατί η κυβέρνησή σας δεν σταμάτησε το σκάφος αυτό που μετέφερε όπλα προς τον δικτάτορα Ασάντ. Για την Τουρκία τώρα. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βότσον ότι οι Τούρκοι πρέπει να σεβαστούν την Προεδρία. Διαρωτώ όμως αν η χώρα σας γνωρίζοντας τις θέσεις που έχει απέναντι στην Τουρκία και το ότι ένα τμήμα της χώρας σας κατέχεται από τουρκικές δυνάμεις, ε, έχοντας όλα αυτά υπόψη, μήπως ε, θα μπορούσατε να κάνετε ένα βήμα να εκπλήξετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σαν παράδειγμα και την Τουρκία ανοίγοντας τα κεφάλαια 23 και 24. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για σας αλλά αυτό θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα και αυτό θα έφετε την Τουρκία μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός. Για το κοσυφοπέδιο τώρα. Άκουσα αυτά που είπατε ότι θα είσαστε επικοδομητικοί και πραγματίστρια. Γνωρίζω ότι η Κύπρος δεν έθεσε βέτο, τελειώνω πρόεδρε, την μελέτη για μια συμφωνία SAA. Αν πάει καλά η μελέτη αυτή για το εφικτό της συμφωνίας, τότε η Κυπριακή Προεδρία θα επιτρέψει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Κοζάκο Μαρκουλή. Όπως θα γνωρίζει είμαι φίλος της Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια. Το, την Κυριακή μάλιστα στο Λονδίνο θα μιλήσω σε μια συγκέντρωση για το θέμα της, Κυπρια... της τουρκικής κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου. Υπάρχει και το θέμα του μποϊκοτάζ από την Τουρκία της Κυπριακής Προεδρίας. Γνωρίζουμε ότι ζητήσατε και δάνεια από τη Ρωσία τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είναι καθαρά εμπορική αντίδραση μπροστά στην κρίση ή ζητάτε και τίποτε άλλο. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο πρόεδρος Χριστόφιας μας μίλησε για τις κύριες προτεραιότητες την πολιτική το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα όμως το θέμα του Μαυροβουνίου και γενικότερα τι σκοπεύετε να κάνετε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Μάλλον η Κροατία θα είναι η επόμενη χώρα της διεύρυνσης, αλλά θα παίξετε ρόλο καλής θέλησης ε, ε καλής και για το θέμα της Φυρών Μακεδονίας Ξέρω ότι κύριο αρμόδιος είναι ο ΙΕ, αλλά ίσως θα μπορούσατε και εσείς να διαμεσολαβήσετε μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων για να βρεθεί μια λύση στο θέμα της ονομασίας. Και ως φίλος και της Κύπρου και του Ισραήλ χαίρομαι ιδιαίτερα για τις φιλικές σας σχέσεις, αλλά τώρα που ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα αερίου, επειδή είστε και φίλοι χώρα με τους Άραβες και τους Παλαιστινίους, θεωρείτε ότι μήπως θα μπορούσατε να παίξετε ρόλο καλή θέληση και για να συνεννοηθούν οι Άραβες με τους Παλαιστινίους και με το Ισραήλ. Ίσως να υπάρξει περίπτωση στη Συρία μεγάλης εξόδου χριστιανών ιδίω προσφύγων. Εάν η κατάσταση γενικευτεί σε εμφύλιο πόλεμο ή αν υπάρξουν διώξεις από σαλαφιστές η Κύπρος θα πρέπει μάλλον να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα. Πώς το βλέπετε αυτό και μήπως θα μπορούσατε και εσείς να παίξετε ένα ρόλο στη σταθεροποίηση των κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας τόσο ατομικά όσο και σας, σαν εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδος της EFD. Βεβαίως είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο χαρακτήρας της εξάμεινης εκπεριτροπής προεδρίας είναι συμβολικός. Αποδεικνύει ότι στην Ένωση αυτή έχουμε αναπτύξει το αίσθημα της δημοκρατίας και το αίσθημα της δημοκρατίας έχει βάσει κυρίως την ευγένεια. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το αίσθημα της ευγένεια και σε άλλα κράτη της περιοχής για να αντιμετωπίσουν ε, την πραγματικότητα της οικουμενικότητας αλλά και της ίδιας της Κύπρου με την ευγένεια που χρειάζεται η οποία δεν επιδεικνύεται εδώ και 37 και 38 χρόνια με ιδιαίτερη επεσήμανση θα ήθελα να κάνω στον άξονα Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και να σημειώσω ότι προσβλέπω σαν ενεργειακή αγωγή να περάσουν από αυτές τις περιοχές και από αυτά τα κράτη. Ε, Ιδιαίτερως επισημαίνω τις καλές σας σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και προσβλέπουμε ότι οι καλές αυτές σχέσεις θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις αποφασιστικότερου ρόλου και ίσως στην παρούσα φάση αποφασιστικότερου ρόλου από οποιοδήποτε άλλο κράτος στην μεσολάβηση και στην διαχείριση της κρίσεως που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ σοβαρή και επισημένο κυρίως αποτελέσματα της ε, λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης τα οποία ακόμη δεν είναι ορατά και ιδιαίτερα αποτελέσματα σε σχέση με το Συριακό πρόβλημα το οποίο αυτές τις μέρες είναι σε ιδιαίτερη έξαση. Άκουσα με προσοχή τις προτεραιότητές σας ε, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Δεν θα ήθελα όμως να επαναλάβω όσα οι προηγηθέντες ε, συναδελφοί μου ε, επεσήμαναν και ερώτησαν. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι τον ιδιαίτερο ρόλο τον οποίο έχετε σαν Προεδρία σε μια παγκόσμια και πανευρωπαϊκή οικονομική κρίση η οποία τώρα λαμβάνει τον χαρακτήρα της ε, ε, κατά κάποιο τρόπο τελικής φάσης με το τραπεζικό σύστημα να τίθεται υπό κάποιο έλεγχο. Παρακαλώ να μου πείτε ποιες είναι θέσεις σας στο θέμα της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλαβράκο, κύριο Μαυρονικόλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την Υπουργό Εξωτερικών τη Κυπριακή Δημοκρατία, και νομίζω ότι όλη η αναφορά και όλη η τοποθέτηση έχει αγγίξει όλε τι τυχές τη γενικότερη εξωτερική πολιτική που επηρεάζει σήμερα και την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το παγκόσμιο. Θα ήθελα απλώς σαν υποσημείωση να τονίσω ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας έρχεται γεωγραφικά να αναδείξει μείζωνα προβλήματα της περιοχής και να αντιληφθούμε ότι το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κάπως διαφορετικό σε ό,τι αφορά τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι γειτονικέ χώρες. Αγγίξατε πολύ ορθά το θέμα του Παλαιστινιακού, το θέμα της Αραβικής Άνοιξης, το θέμα της Συρίας όπου οι σφαγές συνεχίζονται μέχρι τώρα και πολύ περισσότερο θέλετε να αναδείξετε την δυνατότητα η Κυπριακή Δημοκρατία να συμβάλλει κάπως περισσότερον από άλλες πιθανές χώρες λόγω των καλών σχέσεων και με τον αραβικό κόσμο αλλά και με το Ισραήλ. Θα είναι ευχή έργο αν μπορούσαμε να αναδείξουμε κάποιε συγκεκριμένε πράξει και ενέργειε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία που να αγγίξουν αυτές τις, αυτά τα προβλήματα που είναι και πολύπλευρα και ακούντο σημαντικά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρατε το μεταναστευτικό ρεύμα. Μια άλλη μεγάλη και τεράστια πληγή για ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται αυτό το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, ιδιαίτερα από μικρές χώρες, από κράτη-μέλη της Ένωσης όπως είναι η Κύπρος που είναι νησιά. Και ένα τελευταίο, θα ήθελα να αντιληφθώ την δική σας σκέψη πώς μέσα από την οργανωμένη προσπάθεια και αλληλοκάλυψη με το τμήμα εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της κυρίας Άστον, πώς μπορεί και η Κύπρο να συμβάλλει ούτως ώστε ακριβώς μετά από αυτό το εξάμεινο της Προεδρίας να υπάρξει μια δυνατότητα περισσότερης κοινή εξωτερικής πολιτικής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η κυρία Άστο στο τέλος της ημέρας να μπορεί να μιλά εξ όλων. Ευχαριστώ. Eh, eh, Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, έχω την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και ότι θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρετε θαυμάσια γιατί έχω εμπιστοσύνη και στις ικανότητες σας και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ήθελα μόνο να σας ρωτήσω, βλέποντας την ελεηνή στάση την οποία τηρεί η Τουρκία έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμη και σε αυτό που είπε η κυρία Λούνατσεκ προηγουμένως, να ανοίξουμε δύο κεφάλαια. Ήδη έχει απαντήσει ο κύριος Μπαΐς ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε αποδεκτό και θα δούμε από εκεί και πέρα, από τον Φεβρουάριο και πέρα και γνωρίζοντας όλοι ότι η πατρίδα μας, η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, τελεί υποκατοχή και μάλιστα άγρια κατοχή. Πώς θα συμπεριφερθείτε σε αυτό το διάστημα στις μικρές και μεγαλύτερες προβοκάτσιες που εκδηλώνονται καθημερινά εναντίον της Προεδρίας, όχι μόνο εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δείτε για παράδειγμα το περιοδικό ε, The Parliamentarian που κυκλοφόρησε σήμερα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που θα γίνει όταν αύριο θα πάμε με τη μειχτή Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κωνσταντινούπολη να συνομιλήσουμε. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Θα παρίσταται ή δεν θα παρίσταται η Προεδρία. Θα αρνηθούν να δεχθούν την Κυπριακή Προεδρία. Όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα θα πρέπει να τα ξέρουμε και εσείς θα πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε και εμείς αναμένουμε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γι... γιατί αν δεν συμμορφωθεί η Τουρκία θα πρέπει να διακοπεί πάρα αυτά οποιαδήποτε επικοινωνία με αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε, κύριε Θεοχάρης, ο κύριος Πίκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να υποστηρίξω την εστίαση που έχετε για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την στενή συνεργασία με την κυβέρνηση της Κροατίας για τα υπόλοιπα τμήματα που πρέπει να επιληθούν μέχρι την ένταξή μας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου. Βέβαια η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορία διευρύσεων και είναι η παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πραγματική ασφαλιστική, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι μια χώρα θα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρος ότι και η Κροατία θα συμβάλλει στην πολιτική του να παροτρύνει τις χώρες που είναι εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι οι γειτονές μας να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και να βγουν από το παρελθόν κοινωνικών προβλημάτων και δικτατοριών. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη δύσκολη Προεδρία σας. Ε, Ευχαριστώ. Ο κ. Χατζηγεωργίου τέλος. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. σα καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να μα πείτε αν έχετε την καλοσύνη πώς σχολιάζετε την δήλωση του κυρίου Μπαγίς η οποία έγινε στη Μιχτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκίας ότι αν κατά τη διάρκεια της Προεδρία τη Κυπριακής επιχειρηθεί να ανοιχθούν οποιαδήποτε κεφάλαια η Τουρκία δεν θα συγκατανεύσει πώς ε, αντιμετωπίζετε ή πώς σχολιάζετε τις επανειλημμένες, ίσως ξεπερνούν τις 100 ε, δηλώσεις του κυρίου Μπαγής ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Προεδρία και δεν θα έχει καμιά επαφή μαζί της κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Πώς σχολιάζετε την τοποθέτηση ότι ουσιαστικά η Τουρκία θα εξακολουθήσει κατά αυτή την εξαμηνία να έχει επαφές με την Κομισιόν και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς κατά την άποψή σας εν ώψη αυτής της στάσης της Τουρκίας απέναντι στην Κυπριακή Προεδρία θα πρέπει να αντιδράσουν η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Και το τρίτο, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί η Κύπρος, ένα κράτος του οποίου το 1 τρίτο των εδαφών του κατέχεται από χώρα η οποία αιτείται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν κράτος από τα πιο μικρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν υπήρχε η Μάλτα ίσως το πιο μικρό, ε, με πληθυσμό το 1 τέταρτο του Βερολίνου, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί παίρνει τη θέση ότι κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου ε, δεν θα βάλει καθόλου το Κυπριακό στην ατζέντα. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί τα υπόλοιπα 26 κράτη ε, αν θα κρατήσουν την ίδια στάση. Θεωρώ δηλαδή ότι ενώ είναι σωστή και εκφράζει έναν απίστευτο ρεαλισμό, πατριωτικό ρεαλισμό αυτή η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαρωτούμε ποια ε, είναι η στάση των υπολείπων και αν κατά την κρίση σας ε, οι υπόλοιποι καλά κάνουν να, να συγκρατηθούν πάνω στην ίδια γραμμή ή θα έπρεπε να αξιοποιηθεί η συγκυρία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κλείσει το γύρο των αγορητών. Κυρία Υπουργέ, ε, στο πρόγραμμα προβλέπονται 15 λεπτά για την ε, απάντησή σας. Ελπίζω θα μπορέσετε να περιοριστείτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερη και να καλύψω ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τον γύρο αυτών. πολλές ερωτήσεις αφορούσαν την Αραβική Άνοιξη, τη Συρία, την Αίγυπτο. και γενικότερα τις ιστορικές αυτές, αν μπορεί κανείς να πει, αλλαγές στην νότια γειτονιά μας. Πρόκειται για αλλαγές που κανείς δεν ανέμενε πριν από δύο χρόνια. Δεν υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε περίπτωση οι δικτατορίες αυτές, τα αυταρχικά αυτά καθεστώτα που είχαν διαρκέσει δεκαετίες ολόκληρες, που καταπίεζαν τους λαούς τους για δεκαετίες να μπορούσαν κάποια μέρα να ανατραπούν από άοπλους νέους και νέες στις χώρες αυτές. Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στους λαούς αυτούς, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι θα βρισκόμαστε στο πλευρό τους στον αγώνα αυτών για την αλλαγή μαζί τους στον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό και στον αγώνα για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για κίνους και τις μελλοντικέ γενιές των πολιτών των χωρών αυτών. Γι' αυτόν τον λόγο η Κυπριακή Προεδρία έχει ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες της την νότια διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις αυτές της λεγόμενης, των λεγόμενων χωρών της Αραβικής Άνοιξης. Με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της καταφέραμε να πείσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να οργανώσουν την δεύτερη υπουργική συνάντηση Ένωσης Αραβικού Συνδέσμου υπό την Προεδρία μας. Νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ επίκαιρο και σημαντικό. Εκεί θα συζητήσουμε όχι μόνο αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα για να θεσμοποιήσουμε τις σχέσεις μας περισσότερο με τον αραβικό κόσμο. Είχα μακροσκελή συζητήσεις με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, τον κύριο Λάραμπη, που πρόσφατα είχε έρθει στην Κύπρο και συζήτησα επίσης με την υπάτη εκπρόσωπο την Βαρονέσα Άστον. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η συνάντηση αυτή θα γίνει υπό την Προεδρία μας. Για τη Συρία τώρα. Αυτά που γίνονται στη γειτονική μας αυτήν χώρα, και εδώ προσθέτω ότι οι ακτές της Συρίας απέχουν μόνο 100 χιλιόμετρα από τις δικές μας, τόσο κοντά βρισκόμαστε, ανησυχούμε ιδιαίτερα νιώθουμε βέβαια αποτροπιασμό για τις σφαγές και τον απάνθρωπο τρόπο, την απάνθρωπη συμπεριφορά των αόπλων πολιτών, τις απώλειες ζωών και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώνονται στη χώρα αυτή. Γι' αυτό υποστηρίξαμε από την αρχή τις πρωτοβουλίες του Αραβικού Συνδέσμου και του ΟΗΕ για έναν όσο το δυνατόν συντομότερο μια όσο το δυνατόν συντομότερη λύση για να περάσουν τα πράγματα σε άλλη κατάσταση, για να γίνει μια μετάβαση, διότι είναι προφανές ότι χρειάζεται αλλαγή στη Συρία. Υποστηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία του Κόφι του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου και μας ενθαρρύνει πρόσφατη συνάντηση στη Γενέβη. Θεωρούμε σημαντικό η Ρωσία και η Κίνα να συμμετέχουν και αυτές σε τέτοιες συναντήσεις και έτσι απαντώ μερικώς τουλάχιστον στο ερώτημα τι θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος για να πείσει τη Ρωσία να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τη Συρία. Έχουμε βέβαια διμερείς σχέσεις και συζητήσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία και μακρά φιλία με εκείνην, αλλά θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πάτη εκπρόσωπος, αλλά και ο ΙΕ, ήδη έχουν πείσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να συμμετάσχει και γι' αυτό είχαμε τις θετικές εκείνες εξελίξεις στη συνάντηση της Γενέβης. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί χωρίς τη Ρωσία και την Κίνα μάλλον δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν τα ποθούμενα στη Συρία. Είναι λοιπόν θετικές αυτές οι εξελίξεις, αν και ακόμα χρειάζεται να δούμε αν θα εφαρμοστούν αυτά που υπόθηκαν στη Γενέβη και φυσικά ως Προεδρία εμείς θα συνεργαστούμε στενά με την Κάθριν Άστον, την υπάτη εκπρόσωπο, για να δούμε πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η Κύπρος. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την υπάτη εκπρόσωπο, όχι μόνο για τη Συρία αλλά και για όλη τη, όλα τα γειτονικά μας κράτη και δεσμεύτηκα ως εκπρόσωπος της Προεδρίας να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω παίζοντας το δικό της ρόλο όποτε δεν θα μπορούσε εκείνη σε επισκέψεις στην περιοχή ή σε άλλες δραστηριότητες. Για τη Συρία πάλι ανησυχούμε ιδιαίτερα και γι' αυτό ήδη προσπαθούμε με τέρους μας μέσα στην Ένωση αλλά και εκτός αυτής για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει παράπλευρα για την περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ή για την εκένωση χιλιάδων πολιτών της Ένωσης μπορεί να χρειαστεί να σημειωθεί από τη Συρία αλλά και πρόσφυγες από τη Συρία αλλά και από το Λίβανο. Πρέπει να δοθεί το μήνυμα σωστά ότι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι τουλάχιστον η θέση του Συμβουλίου Εξωτερικών, Υπουργών Εξωτερικών, κανείς στην Ένωση δεν θέλει στρατιωτική παρέμβαση στη Συρία. Αλλά και για την περίπτωση αυτή, την ακραία, που θα υπάρξει εκεί σύραξη, ετοιμαζόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά θα υπάρξουν επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή και οι πρώτοι που θα πληγούν από μια τέτοια, σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι ο γειτονικό μας Λίβανος. Με το Λίβανο επίσης έχουμε πάρα πολύ στενές και πολύ ισχυρή φιλία, σχέσεις και φιλία και δεν θα θέλαμε η χώρα αυτή που έχει υποφέρει τόσο πολύ να καταστραφεί εκ νέου ή να πληγεί εκ νέου. Σε αυτά τα σχέδια λοιπόν για πιθανή εκένωση μέχρι 100.000 πολιτών της Ένωσης και πολιτών τρίτων χωρών ετοιμαζόμαστε. Επίσης υπόθηκαν πολλά για την Τουρκία και την ατυχή στάση που τηρεί η τουρκική δημοκρατία ως προς την Προεδρία μας. Λέω ατυχή διότι το λέω ευγενικά. Γιατί πρόκειται για χώρα που στοχεύει στην ένταξή της στην οικογένεια αυτή εθνών. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη χώρα που να είναι υποψήφια για ένταξη στην Ένωση και να φέρεται προς μια ήδη χώρα μέλος με τέτοιον τρόπο απαράδεκτο. Λέγοντας δηλαδή ανοιχτά ότι δεν αναγνωρίζει τη χώρα αυτή, ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν τρόπο με την Προεδρία και μάλιστα να τα καταφέρνει κιόλα. Αυτό για μας είναι αδιανόητο ότι μπορεί να συμβεί, ότι θα μπορούσε να συμβεί και όμως συνέβη αλλά όπως είπα και προηγουμένως θα ακολουθήσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με ρεαλισμό είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με την Κομισιόν και με την Τουρκία εάν και εφόσον η Τουρκία αποφασίσει και εκείνη να συνεργαστεί με την Προεδρία. Όπως όμως είπαμε ήδη και το επαναλαμβάνω, ο κύριος Μπαγής, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, ήδη αποσαφήνισε ότι δεν θα συνεργαστεί η Τουρκία ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματο νέων κεφαλαίων στις συνταξιακές διαπραγματεύσεις. Ούτε τότε θα συνεργαστούν κατά την εξάμηνη αυτή περίοδο της Προεδρίας μας. Αυτό το είπαν καθαρά. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία πιθανότητα να το αμφισβητήσουμε αυτό ή να φανταστούμε άλλα σενάρια. Για να είμαι ειλικρινής βέβαια εμείς θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν η Τουρκία άλλαζε τη στάση της και συνεργαζόταν με την Κυπριακή Προεδρία. Τότε θα βλέπαμε τι, μπορούσε θα μπορούσε να γίνει. Όπως ξέρετε υπάρχουν τρία κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Η Τουρκία δεν ζήτησε το άνοιγμά τους και εμείς με τα χαρά θα συνεργαζόμασταν και με την Τουρκία και με την Κομισιόν για να ανοίξουν τα κεφάλαια αυτά, τα τρία αυτά κεφάλαια. Για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι ατυχές που δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με τη ΦΥΡΟΜ εγώ τελευταία ανέλαβα μια πρωτοβουλία γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη μια τέτοια κατάσταση να μην έχουμε διπλωματικές σχέσεις δηλαδή με μια υποψήφια χώρα. Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία, συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών της ΦΥΡΟΜ και πρότεινα ορισμένους τρόπους για την δημιουργία διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά μέχρι σήμερα δεν είχα ανταπόκριση. Επειδή όμως είμαι επίμονη και θα επανέλθω, σύντομα θα ξανασυναντηθώ με τον Υπουργό Εξωτερικών και είμαι βέβαιη ότι αν υπάρχει καλή θέληση θα υπάρξει και ο τρόπος να γεφυρωθεί αυτό το κενό, γιατί είναι κενό που δεν έχουν σχέσεις διπλωματικές οι δύο μας χώρες. Uh, to Mr. Uh, Watson. Προς τον κύριο Watson θα ήθελα να πω ότι δεν κατάλαβα καλά το σχόλιο σας ότι δηλαδή η διέρεση της χώρας υπονομεύει την αξιοπιστία της Προεδρίας. Είμαι βέβαιη κύριε Γουάτσον ότι γνωρίζετε Α, συγγνώμη, δεν σας έβρισκα. Τώρα ήρθατε μόλις ακούσατε το όνομά σας. Τι έγινε. Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε τις προσπάθειες της Κυπριακής κυβέρνησης και της ελληνοκυπριακής κοινότητας κατά την 38 ετή αυτή περίοδο για επανένωση της χώρας. Παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα, ο κυριότερος στόχος μας να ενωθεί η χώρα. Η... Ο διαχωρισμός, η διέρεση δεν είναι μόνο κάτι απαράδεκτο, ο διχασμός, αλλά και ένα μια πληγή στο σώμα της Κύπρου και στην ψυχή της Κύπρου. Πρέπει να επανενωθεί η χώρα. Αλλά θέλουμε ακριβώς αυτό, ένωση της χώρας ομοσπονδιακή, όχι συνομοσπονδιακή με δύο χωριστές χώρες. Και γι' αυτό δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να συμφωνήσουμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν με αυτή την έννοια μπήκαμε και στην Ένωση το 2004 με την έννοια ότι όλη η Κυπριακή επικράτεια όπως γνωρίζετε καλά έχει ενταχθεί εκτός από τις δύο κυρίαρχες βάσεις. Το σύνολο της νήσου έχει ενταχθεί Αυτό το δέχτηκε και η Βρετανία κατέχει τις δύο κυρίαρχες βάσεις. Πάντως ο στόχος μας είναι η επανένωση της χώρας και θα συνεχίσει να είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Όσο για την ε, Partnership for Peace, έχετε εσείς κανένα καλύτερο νέο από την Τουρκία κύριε Βάτσον. Δηλαδή, αν κάνουν την αίτηση θα το υποστηρίξετε. Αν ναι θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα γιατί ξέρετε ότι η Τουρκία μπλοκάρει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πάνω από 20 διεθνείς οργανώσεις, ασκή, άρνηση κυρία και βέτο. Και φαντάζομαι το ίδιο θα κάνουν και για αυτό το θέμα. over these past uh, few weeks and uh, months. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες νομίζω ότι η θέση μας υπήρξε σαφής ως προς το πλοίο. Ξέρω καλά τι έγινε και θα ήθελα να σας εξηγήσω και σε εσά και στα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου υπό ποιε συνθήκες συνέβη το περιστατικό. Το πλοίο αυτό που ήταν ρωσικό με σημαία Γρεναδίνων έφυγε από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό το Ισκεντερούν την Αλεξανδρέτα. Ο προορισμός από την αρχή του ταξιδιού ήταν το Ισκεντερούν. Το πλοίο πλησίασε την Κύπρο, δεν μπήκε στα χωρικά ύδατα, δεν μπήκε στο λιμάνι της Λεμεσού. Παρέμενε έξω από το λιμάνι, υπήρχε κακοκαιρία και ζήτησε ανεφοδιασμό. Δεν μπορούσαμε να τον αρνηθούμε και ανεφοδιάσαμε το πλοίο σε καύσιμα. Όταν όμως ελέγξαμε τα χαρτιά του, φάνηκε ο προορισμός που ήταν το Ισκεντερούν και μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις και από τον πλοίαρχο και από τους ιδιοκτήτες και από την εταιρεία που διαχειριζόταν το πλοίο στη Λεμεσό ότι ο προορισμός του θα ήταν το Ισκεντερούν και γι' αυτόν τον λόγο του επιτρέψαμε να αποχωρήσει. Δυστυχώς όμως αντί για Ισκεντερούν το πλοίο πήγε αλλού στο Ταρτού, στην Ταρτισό της Συρίας. Πρέπει να σας πω ότι η Κυπριακή κυβέρνηση προσέφυγε ποινικά κατά του πλοιάρχου της εταιρείας ρωσικής εταιρείας στην οποία ανήκει το πλοίο και κατά της διαχειριστικής εταιρείας στη, στη Λεμεσό, στην Κύπρο. Και η προσφυγή αυτή είναι στα κυπριακά δικαστήρια. Αυτό θέλω να το γνωρίζετε. Η κυπριακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας εφαρμόζει πλήρως τη διεθνή νομοθεσία και τις κυρώσεις. Πέρυσι, όπως ξέρετε, με το θάνατο 13 νέων πληρώσαμε βαρύ τίμημα. Καταστράφηκε όπως γνωρίζετε η ηλεκτρική υποδομή μας διότι ακριβώς εφαρμόζουμε τις κυρώσεις και γιατί κατασχέσαμε ένα πλοίο το 9 που μετέφερε παράνομα όπλα στη Συρία. Αυτό ήθελα να το ξέρετε και ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό. Πάλι για τον κύριο Μπαγής νομίζω το είπα. Το είπα. Τώρα για την τουρκική κατοχή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβουμε πράγματα που έχουμε ξαναπεί, που είπε προηγουμένως κυρία Θεοχάρους. Είναι κατάσταση που τη γνωρίζει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια σαφής θέση από τα πολλά ψηφίσματα που έχει εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ΙΕ. Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ τώρα. και τη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Θέλω να κάνω σαφές ότι, <clears throat> ότι η Κύπρος και η αντιμετώπιση της Κύπρου είναι ότι πρέπει να συνεργάζεται με όλους τους γείτονές της. Ιδίως στο νέο αυτό γεωγραφικό χώρο συνεργασίας που συμπεριλαμβάνει και την ανακάλυψη και εκμεταλλεύση θράκων. Βάσει εκτιμήσεων από τη Γεωγραφική, Γεωλογική Εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών καλύπτει 453 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ε, φυσικού αερίου και 10 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής και γι' αυτό η Δημοκρατία της Κύπρου έχει ξεκινήσει ενέργειες συνεργασίας με όλους τους γείτονές της <clears throat> για να μπορέσουν να δημιουργήσουν από κοινού το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία αυτού του είδους. Συνεργασόμαστε με το Ισραήλ, συνεργασόμαστε με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο και φυσικά υπάρχει περιθώριο πάντα για συνεργασία με την Τουρκία στο μέλλον, εφόσον η Τουρκία φυσικά επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου και την υπέρβαση του κυπριακού προβλήματος και στοχεύσει στα πραγματικά ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Τουρκία, ο λαός της και όλη αυτή η περιοχή μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας και ειρήνης που θα αποβεί προς το καλό όλων των χωρών της περιοχής. Αυτό είναι το όραμά μας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον. <clears throat> Υπάρχουν επίσης και άλλοι τομείς συνεργασίας <clears throat> με τις χώρες της περιοχής, περιοχής. Μία από αυτές είναι η σύνδεση του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος και μέσω της Ελλάδος την σύνδεση με την Ευρώπη με ηλεκτρικό καλώδιο, με ηλεκτρικό δίκτυο αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας, εφικτού και αυτός μπορεί να είναι ένας νέος χώρος συνεργασίας. Συγχρόνως όμως προχωρούμε και σε συνεργασία με τους άλλους γείτονές μας στον αραβικό κόσμο. Πιστεύω λοιπόν ότι έχω γενικά καλύψει τα ερωτήματά σας. Ζητώ συγγνώμη και απολογούμε αν κάποια τα ξέχασα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαρκουλή, κυρία Υπουργή, Υπουργέ. Όπως ε, είπαν και οι συναδελφοί μου, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εξαμηνία Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ και πάλι και ξαναδίνω την Προεδρία στον κύριο Μπρόκ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με το σημείο 21. Σύσταση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη νέα Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Ο κύριος Βόμποντα έχει το λόγο, αν δεν ενοχλεί τις ωραίε κυρίες. Ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος προηγείται, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Συνάδελφοι, σύντομα θα παρουσιάσω την έκθεσή μου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, την έχετε την έκθεση γραπτά. Να ξεκινήσω με τις βασικές γραμμές. Απαιτείται μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να ασκούμε κριτική σε κάποια από τα χαρακτηριστικά της Ρωσίας. Η ελπίδα μας ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά, χρόνο με το χρόνο διαψεύδεται. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, να ασκήσουμε πιο αυστηρή κριτική από ό,τι θα θέλαμε με έναν εταίρο. Να μιλήσω λίγο για τα χαρακτηριστικά της εταιρικής αυτής σχέσης. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είναι στρατηγική σχέση ή όχι. Θα έπρεπε να είναι στρατηγική η σχέση αυτή. Αλλά οι, οι προϋποθέσεις για να γίνει η Ρωσία στρατηγικός εταίρος δεν έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί ένα στρατηγικός εταίρος θα πρέπει ένας εταίρος με τον οποίο να έχει κανείς πολλά κοινά, κοινούς στόχους, θα πρέπει να προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια κάποια διατύπωση η οποία θα καταστήσει τη Ρωσία στρατηγικό εταίρο, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν έχουν εκπληρωθεί θα έλεγα. Τώρα για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά οι επαφές μου με την διαπραγματευτική ομάδα είναι ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, αλλά η πρόοδος είναι μικρή και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι δημοκρατικές αρχές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή. Η σχέση μας με τη Ρωσία δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο οικονομικές πλευρές. Αυτό είναι σαφές. Και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα αργότερα διευκρινίζοντας ότι αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει με τον νόμο για τις ΜΚΟ είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολλές αμφιβολίες. Βέβαια οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ πρόσφατες και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση μία θα έλεγα αξιολόγηση και κριτική του συγκεκριμένου νόμου. Η ιδιότητα του μέλους στον ΠΟΕ είναι κάτι το οποίο δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τη Ρωσία και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Η Ρωσία επανειλημμένα λέει ότι έχουμε μια τελωνιακή ένωση οπότε η σχέση μας εντάσσεται στα πλαίσια της τελωνιακής αυτής ένωσης. Αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος. Εμείς διαπραγματευθήκαμε με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτή τη διαπραγμάτευση. Σε μια δεύτερη φάση μπορούμε να μιλήσουμε ε, για την Τελωνιακή Ένωση, αλλά προς το παρόν μιλάμε με τη Ρωσία και όχι με την Τελωνιακή Ένωση, μια άλλη οντότητα. Κάτι τέτοιο δεν θα είχε πάρα πολύ μεγάλο νόημα για μας. και δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να πιέσουμε την Ουκρανία και μόνο. Για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία αναφέρθηκα ήδη στην κοινωνία των πολιτών, στην έλλειψη μεταρρυθμίσεων και θα πρέπει να αναφέρουμε το θέμα της νέας νομοθεσίας, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα δυστυχώς στην κοινωνία των πολιτών. Τους τελευταίους μήνες δημιουργούνται πιέσεις προς την κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώς δεν στηρίζεται επαρκώς από τον πληθυσμό η πλευρά αυτή της ρωσικής κοινωνίας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία και σε σχέση με τις ενέργειες της κυρίας Σόπτσακ να δούμε τι θα κάνει η αστυνομία αν συνεχίζει να μπαίνει σε σπίτια για έρευνες, να δεσμεύει χρήματα κτλ. Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχει και το θέμα ενίσχυσης του διαλόγου με την ε, Ρωσία. Επανειλημμένα ακούμε εμείς τη δικαιολογία ότι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν και σε ευρωπαϊκές χώρες. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ ψάχνουμε το τι γίνεται στη Ρωσία. Και μπορούμε να ακούμε τις ιδέες τους, να υφιστάμεθα την κριτική τους, αλλά βασικά η δυνατότητα θα πρέπει να είναι από πλευρά μας να ακούγεται η άποψή μας. Η διαφθορά είναι κάτι το οποίο προανέφερα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσει η Ρωσία προς το δικό της συμφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια για τις επενδύσεις λόγω της διαφθοράς. Δεν ξέρω ότι οι επιχειρήσεις δεν επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή. Η διαφθορά δεν είναι μόνο κεντρική κρατική, αλλά εξαρτάται επίσης και από τις τοπικές αρχές, από τις περιφερειακές αρχές και είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Για τις διεθνείς προκλήσεις είναι σαφές το τι θα πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι και η οικονομία βέβαια και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Αυτό δεν είναι κάτι το αυστήρα τεχνικό οικονομικό. Αυτό περιλαμβάνει και το σεβασμό του κράτους δικαίου, μια κοινωνία ανοιχτή και σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων. Έχει σημασία λοιπόν να υπάρχει μια συνολική αντίληψη για το τι σημαίνει μια οικονομία έχει σημασία λοιπόν αυτό για μας η ενέργεια, η συνεργασία στον κλάδο της ενέργειας είναι καθοριστική, αλλά εμείς θα πρέπει να αποφασίζουμε για το από πού θα αγοράζουμε ενέργεια. Είναι σαφές ότι η Ρωσία θα παραμείνει για πολλά χρόνια σημαντικός παράγων στον τομέα της ενέργειας και, της, και των πηγών παραγωγής ενέργειας. Το θέμα θα μείνει στην ημερήσια διάταξη γιατί ο διάλογος με τη Ρωσία θα είναι πιο δεκτικός, πιο παραγωγικός, πιο ανοιχτός εφόσον και εμείς επιλέγουμε τα θέματα τα οποία θα συζητάμε μαζί τους. Λοιπόν, για την, έχουμε την έκθεση για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια. Θέλουμε μια στενή εταιρική σχέση, θέλουμε η Ρωσία να είναι στρατηγικός εταίρος, αλλά θα πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να γίνουν μεταρρυθμίσεις μέσα στη Ρωσία, γιατί δεν βλέπουμε πραγματική πρόοδο μέχρι τώρα. Και τα θέματα που έχουν σχέση με τη Ρωσία δεν θα πρέπει να αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί να υπάρξει εταιρική σχέση Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχουν νόμοι για ΜΚΟ, που εμποδίζουν τις ΜΚΟ να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. και ευρωπαϊκές ε, ΜΚΟ και ΜΚΟ από τη Ρωσία δυσκολεύονται να δουλέψουν σοβαρά και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Έχουν γίνει προσπάθειες, οι προσπάθειες αυτές δεν ήσαν ικανοποιητικές μέχρι τώρα. Θα πρέπει οι Ρώσοι να δείξουν σεβασμό όχι μόνο στην κοινωνία των πολιτών τους, αλλά και στις ΜΚΟ τους που παλεύουν για αλλαγές στη Ρωσία. Η έκθεση συνολικά δεν χαρακτηρίζεται σαν θετική λοιπόν, αλλά από ό,τι μαθαίνω από τους διαπραγματευτές βρισκόμαστε στο πρόωρο ακόμα στάδιο. Είμαι θετικός σε σχέση με μέτρα όπως η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, αλλά η ανταπόκριση από τη Ρωσία μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαιτέρως πιστική. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική ισορροπία. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να κάνω την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Σφόμποντα. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν ως κοιόδηση συγγήτρια από το ΕΛΚΑ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ευχαριστία μου στον κύριο Σφόμποτα για την, για την πρόταση του ψηφίσματος. Νομίζω ότι είναι πλήρης και πολύ θετική αυτή η διατύπωση που έχει ακολουθήσει. Και συμφωνώ και με το περιεχόμενό της. Η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το κείμενο αυτό σύντομο με μια καλή συνεργασία μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών, σκιωδών εισηγητών. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι πια καιρός να δημιουργήσουμε ένα συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουν λάβει χώρα πολλά σε αυτήν την συνεργασία, τα οποία δεν ήταν πάντα θετικά. Πιστεύω λοιπόν ότι η στρατηγική αυτή εταιρική σχέση την οποία θέλουμε να οικοδομήσουμε θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια νέα συνθήκη, με μια νέα συμφωνία με την Ρωσία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να πούμε ότι εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς, δεν έχει νόημα να έχουμε μια νέα συνθήκη. Μια νέα συνθήκη θα πρέπει να είναι στραμμένη προς το μέλλον. Η Ρωσία είναι ένας μεγάλος, σημαντικός γείτονάς μας. Έχουμε μια σημαντική ε, σειρά θεμάτων που μας εμπλέκουν. Γνωρίζω όμως και τους Ρώσους συναδέλφους, εάν θέλουν να τροχοπεδίσουν τη διαδικασία λόγω λεπτομεριών, θα πρέπει να τους πείσουμε ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι να έχουμε μια σύντομη και σαφή συνθήκη η οποία θα γίνει σεβαστή και μια βασική αρχή που πρέπει να διέπτει σχέση μας με τη Ρωσία είναι η αρχή της αμοιβαιότητος. Χωρίς αυτή την αρχή τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Κατανοώ ότι η Ρωσική Δούμα πριν από μία ώρα ενέκρινε τη συμφωνία με τον ΠΟΕ. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και η ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, συμφωνίες πλαίσιο που υπάρχουν με τον ΠΟΕ. Υπάρχουν ε, και θέματα σε σχέση με το τα Κύριε Ασπέργης λέει η ομιλητρία. Έχει διαφορετική ατζέντα ο κύριος ε, Λαντσπέργκης, φαίνεται. Οι συμφωνίες λοιπόν που χρειαζόμαστε στον εμπορικό τομέα και στον οικονομικό τομέα σε λίγο θα πει ότι δεν ε, συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Λαντσπέργκης, αλλά δεν με ακούει λέει η κυρία Όμεν Ράιτεν από την ε, πλευρά της οικονομίας, του εμπορίου και της ενέργειας θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Χρειάζεται να μιλήσουμε και για αξίες δημοκρατικές, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά αν θέλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο. Το είπε και ο κύριος Σφόμποντα. Το θέμα της ενέργειας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και νευραλγικό θέμα αυτό το οποίο με εντυπωσίασε είναι ότι το μανιφέστο για την ενέργεια ε, που ήταν μία από τις προηγούμενες συμφωνίες μας, ότι αυτή η έκφραση δεν αναφέρεται καθόλου στην, ε, στην έκθεσή του. Ορισμένα πράγματα τώρα πιο εξειδικευμένα. Αναφέρατε την έννοια των benchmarks στην συμφωνία αυτή εταιρικής σχέσης και σύνδεσης. Θέλουμε απλώς μια εταιρική σχέση ή θέλουμε και μια σχέση σύνδεσης. Η διμερής λοιπόν αυτή συμφωνία θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Η εταιρική σχέση, η συμφωνία σύνδεσης. Επίσης, η τελωνιακή ένωση. Εγώ τρέφω πολλές αμφιβολίες. Αν η Ρωσία έχει <clears throat> μια τελωνιακή ένωση, παραδείγματος με το Καζακστάν, η Λευκορωσία, αν αυτή η τελωνιακή ένωση θα πρέπει να αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το ξέρω αυτό αν πράγματι έτσι είναι βάσει του κειμένου. Κύριε Σφόμποντα, το κείμενο αναφέρεται επανειλημμένα στις διεθνείς υποχρεώσεις των συμβαλωμένων μερών. Ίσως όμως και η Ρωσία θα πρέπει να αναλάβει περισσότερο τις διεθνείς ευθύνες της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες σύντομες παρατηρήσεις και σε συνεργασία μαζί σας κύριε Σφόποτα θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε καλύτερα το κείμενο, να το προσαρμόσουμε και νομίζω ότι μπορούμε έτσι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα παραμένοντας βέβαια μέσα στα πλαίσια της συντομίας ως ΕΛΚ εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας ώστε το κείμενο αυτό να είναι συγκεκριμένο, σαφές και να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης από το Κοινοβούλιο μας και φυσικά θα οδηγήσει σε μια ταχεία δράση από εμά, γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχουμε χωριστές συμφωνίες με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Κυρία Όιμερ Ρόιτεν, θέλω να υπερασπιστώ καταρχήν το δικαίωμα των μεμονωμένων βουλευτών να κοιμούνται εφόσον το επιθυμούν. κυρία Όουλαντ. Να πω λίγα πράγματα θα ήθελα να πω. Πρόκειται για μια καλή πρόταση, συνολική θα έλεγα πρόταση. δίνει αρκετά στοιχεία τα οποία θα χαρακτηρίζουν τη διμερή μας σχέση με την Ρωσία. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Ρωσία δεν είναι μόνο μία εταίρος, είναι μέλος όμως του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει αναλάβει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όταν εντάχθηκαν σε οργανώσεις διεθνείς και ιδιαίτερα στο Συμβουλίο της Ευρώπης. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, λίγες παρατηρήσεις για την κοινωνία των πολιτών. Αναφερθήκατε στους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία στη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό γίνεται όλο ένα και πιο μεγάλο εμπόδιο για τη Συμφωνία Σύνδεσης ή μάλλον για την ελευθερία στην Ρωσία. Είχαμε εκπροσώπους με τη, της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα προβλημάτων που δημιουργούνται Και η τελευταία προσπάθεια αφορά όχι μόνο την ομοθεσία αλλά και μια σκληρή προπαγάνδα εις βάρος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που κατηγορούνται σαν κατάσκοποι της δύση. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να καταλάβω πως τέτοιου είδους προπαγάνδα εξυπηρετεί συγκεκριμένου στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι που ε, έχουν οι αρχές στο Κρεμλίνο. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για βραχυπρόθεσμα ταξίδια. Οι διευκολύνσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο για τους φοιτητέ, αλλά και τους επιχειρηματίες. Τώρα που εντάσσεται η Ρωσία στον ΠΟΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται η Ρωσία με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης και να μπορέσει να εφαρμόσει ακριβώς όλα αυτά τα σημεία του οδικού χάρτη. Το λέγω αυτό γιατί βλέπω όλο και περισσότερο κάποιους εκπροσώπους της κοινωνίας της επιχειρηματικότητας της Ρωσίας να φεύγουν από τη Ρωσία για να απελευθερωθούν από το καθεστώς εκεί και να μπορέσουν να ταξιδέψουν ελεύθερα συχνά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην χορήγηση των θεωρήσεων είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις και σημαίνει ότι οι διμερείς σχέσεις ακόμα και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Τώρα για τα θέματα της διαφθοράς υπήρξαν συγκεκριμένες αναφορές Σχετικά με την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, θα πω ότι τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε από τους ομολόγους μας, από την κοινωνία των πολιτών, από την αντιπολίτευση, το θέμα της διαφθοράς είναι κάτι το οποίο συνδέεται με το καθεστώς του Κρεμλίνου. Συνεπώς, η είσοδος της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα διευκολύνει όλες αυτές τις διεφαρμένες δομές στην Ρωσία, θα τους διευκολύνει επιχειρηματικά, θα βελτιώσει τις επαφές τους με την Δύση γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε, να γίνουμε ακόμα πιο ξεκάθαροι θα έλεγα Υπάρχει ομάδα Κλουεύ η οποία συνεχίζει να εργάζεται. Παρακολουθεί τις ροές των βρώμικων χρημάτων που κυκλοφορούν ανάμεσα σε διάφορες χώρες, τις απάτες που γίνονται στον τομέα των κατοικιών οικοδομών και κάτι θα πρέπει να γίνει με τα θέματα αυτά γιατί δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον μας να συνεχίσει η κατάσταση αυτή ως έχει και είναι εις βάρος ε, και του ε, μεσαίου Ρώσου πολίτη. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να συνεργαστούμε και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές και νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Κύριε Σούλτς. Είναι πολύ καλό ότι έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης και έχουμε ακούσει και τα σχόλια του εισηγητή, τον οποίο εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα καταλήξουμε και σε ένα καλό κοινό παρονομαστή. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπήρξαν μικρές πρόοδες στη συνεργασία με τη Ρωσία. Αντίθετα πιστεύω ότι υπήρξαν υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις στα θέματα αυτά. Δεν έχουμε στρατηγική συνεργασία αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε ακόμα σε κάποια απόσταση ημένα από τους ΔΕΗ και δεν έχουμε και μία στον τομέα της ασφάλειας συνεργασία. Βλέπουμε στη Συρία να έχουμε μία τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Η, η Ρωσία είναι συνυπεύθυνος και συνένοχος σε αυτήν την κατάσταση και στην καταστροφική στάση που ακολουθεί ο Μπασίρα Λασάντ. Το ίδιο ισχύει και για την ε, διαμάχη μας με το Ιράν. Ούτε και εκεί υπάρχει στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία, ούτε για την αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ. Η ρωσική απάντηση ήταν το να εγκαταστήσει πυράβλους στο Καλίνιγκραντ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά συγκροτούν μία στρατηγική συνεργασία. Απλώς θα πρέπει να κάνουμε αυτά που είναι απαραίτητα για να αποτρέψουμε μια επιστροφή στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δεύτερον, δεν μπορούν να υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας με μια τελωνιακή ένωση. Για τον Πούτιν είναι μια ευρασιακή ένωση. Θέλει πάντα η Ρωσία να έχει μια ιδιαίτερη θέση, δεν θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα της ε, πολιτικής γειτονίες Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά, θέλει να αντιμετωπίσει το υπερδύναμη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως θέλει, είναι ένα από τα παιχνίδια, από τα κόλπα του, του Πούτιν, να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με μια ευρασιατική συμμαχία που περιλαμβάνει και την Λευκορωσία του Λουκασένκο. Είναι όλο αυτό μια προσπάθεια διέρη και βασίλευε που ακολουθεί ο Πούτιν, ο οποίος θέλει να διαπραγματεύεται διμερώς με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι οι φόβοι των ε, αντιφρονούντων τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ότι θα υπάρξει περιορισμός των αστικών ελευθεριών ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Έχουμε τώρα ένα μη νομιμοποιημένο κοινοβούλιο το οποίο επιφέρει περιορισμό του δικαιώματος του συνέρχεστε και ε, μειώνει τις δυνατότητες για διαδηλώσεις. Αυτός ο νόμος βρίσκεται τώρα σε μια πρώτη ανάγνωση. Βλέπετε ότι οι διαδηλωτές ουσιαστικά θα θεωρούνται ως πράκτορες ξένων συμφερόντων και θα σπηλώνονται με τον τρόπο αυτό. Και ίσως καταλαβαίνει ακόμα και η Ντούμα ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια ε, αρνητική αντιμετώπιση για την εικόνα της Ρωσίας στο παρελθόν. Η οργάνωση αυτή Γκόλος που αναφέρθηκε προηγουμένως. Κανονικά αυτό είναι μια ομάδα από ΜΚΟ που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και είναι σημαντικό να έχουν και υποστήριξη από έξω όπως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νόμος για το διαδίκτυο επίσης ο οποίος προβλέπεται να εξεταστεί από τη Δούμα έχει δημιουργηθεί μια, ένας κοινό δημόσιος χώρος στο διαδίκτυο τη στιγμή που τα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία είναι φημωμένα σε μεγάλο βαθμό αλλά με το πρόσχημα μιας νομοθεσίας για την πορονογραφία φαίνεται ότι η έννοια της πορνογραφίας στη Ρωσία είναι ιδιαίτερα ευρεία και έχει σαν στόχο να φημώσει την αντιπολίτευση. Η περίπτωση, της, ε, περίπτωση και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούνται οι αντιφρονούντες είναι εύγλωτος. Βλέπετε ότι ο αρχισυντάκτης Σόκολοφ της Νόβα για έχει ε, απαχθεί και κάποια στιγμή μάλλον απειλήθηκε και με εκτέλεση. Όλα αυτά δείχνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Όπως φάνηκε και από την περίπτωση Μαγνίσκη, υπάρχει αυτή η τρομοκράτηση των αντιφρονούντων και γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να συμμεριστώ αυτή την ιδιαίτερα ροδόχρωα και αισιόδοξη παρουσίαση που έχει γίνει για τη Ρωσία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και τίμοι και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν λέμε ότι βλέπουμε μια θετική εξέλιξη στη Ρωσία, φοβάμαι ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σόμποντα, για το σχέδιο έκθεσής του, το οποίο μας προσκαλεί όλους σε μια γενική εξέταση και προβληματισμό για τα θέματα αυτά. Ε, ελέγχθη σήμερα ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί τόσο γρήγορα μια στρατηγική συμμαχία με την Ρωσία. Και ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε είναι ότι αν δεν πρόκειται να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γιατί όχι. Ίσως θα ήταν χρήσιμο λοιπόν η έκθεση να δίνει κάποιες απαντήσεις στο γιατί όχι. Σε ένα σημείο του ο εισηγητής αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αγγλικά συνεχίζει να είναι προσιλωμένη στην ανάπτυξη και την εμβάθυνση των σχέσεών της με τη Ρωσία επί τη βάση κοινών συμφερόντων και της προσήλωσης της παγκόσμιες αρχές και αξίες. Συμφωνώ με κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι επαρκές να βασιζόμαστε μονάχα σε μια τέτοια διατύπωση. Εμείς, αν θέλουμε να έχουμε μια πλήρη στρατηγική ε, σχέση, αυτή θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να έχει μέλλον. και θα πρέπει να βασιζόμαστε σε κοινέ αξίες για να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια στρατηγική σχέση. Μόνο σε δύο άλλα σημεία, στο σημείο N και στο σημείο O, αναφέρει ο εισηγητής τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε κοινά συμφέροντα. Αναφέρεται στις παγκόσμιες προκλήσεις, στη μη διασπορά πυρηνικών όπλων, στην ε, ειρηνική λύση των ε, συγκρούσεων, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της κλιματικής αλλαγής, μείωση της ένδυας και αναφέρεται κάπου αλλού στην ε, σταθεροποίηση και την πολιτική και οικονομική συνεργασία. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μια σύσταση προς την Κομισιόν, προς το Συμβούλιο, την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Ποια είναι η σύστασή μας σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά να μας οδηγήσουν σε περαιτέρω επεξεργασία από την πλευρά του εισηγητή, να τα εμβαθύνει για να έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία θα διατυπώσουμε υπό μορφή συστάσεων και που να οδηγούν και σε μια πιο συγκεκριμένη σύσταση για την εντολή διαπραγματεύσεων και για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πράγματι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι αυτή που θα περνώ τη συνομιλητής μα και όχι η Τελωνιακή Ένωση στην οποία συμμετέχει η Ρωσία θα πρέπει να κάνουμε σαφές τι περιμένουμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Περιμένουμε να είναι ένας εταίρος διαπραγματεύσεων και να ε, καθορίσει τη στάση της σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι συνεκτικός για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στις μελλοντικές μας σχέσεις και στα κοινά σημεία που θα πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο βλέπω ένα τομέα να λείπει τελείω, που είναι ο πολιτισμός, η επιστήμη, η έρευνα κτλ. Είναι ένα τομέα όπου μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία και εγώ βρίσκω σημαντικό αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Σούλτς, ο οποίος αναφέρθηκε επικριτικά για το σχέδιο του εισηγητή. Όλα αυτά τα οποία αφορούν το, την νομοθεσία για τις ΜΚΟ θα πρέπει και το δικαίωμα του συνέρχεστε θα πρέπει να συμπεριληφθούν γιατί απο, αφορούν και μια κριτική δική μας για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσική Ομοσπονδία αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητο να έχουμε σαφήνεια και διαφάνεια και να εξασφαλίσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ρωσική Ομοσπονδία ότι εμείς υποστηρίζουμε την ανάγκη δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Χαίρομαι λοιπόν με στιγμή για την συνεργασία με τον εισηγητή και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια κοινά σημεία τα οποία θα οδηγήσουν σε μια πλήρη και εξισορροπημένη έκθεση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να είσαστε λίγο πιο σύντομοι, λέει ο πρόεδρος, γιατί έχουμε προβλήματα με την χρήση του χρόνου. Δύο λεπτά σας παρακαλώ. Κρίμα Ήθελα να μακρηγορήσω λίγο περισσότερο. Τι μπορώ να κάνω όμως. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή γιατί έκανε πολύ σημαντική δουλειά ο κύριος Βόμποντα. Εγώ ανέμενα 4-5 χιλιάδες τροπολογίες και του δίνω τα συλληπιτήριά μου αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα στην έκθεση και εγώ θα καταθέσω τροπολογίες να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τη Ρωσία. Γιατί ήμουν και εγώ εισηγήτρια για, το, για την ξυλία και άλλες πρώτες ύλες και γνωρίζω το πρόβλημα, καθώς και για τις απάτες και απομιμήσεις που είναι σημαντικό πρόβλημα στη Ρωσία, καθώς και για την πνευματική ιδιοκτησία. Είναι θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο και άλλα προβλήματα ως προς την προμήθεια ενέργειας στις βαλτικές χώρες, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία. Πρέπει να βιαστώ βέβαια, αλλά Θέλω να προσθέσω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διαφορετική αντίληψη για την ιστορία και θα πρότεινα τη δημιουργία μιας σχετικά μόνιμης ομάδας συζήτησης του θέματος αυτού της ιστορίας. Ας σας πω τώρα δυο λόγια και για τις θεωρήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όπως η συνάδελφος Όιλαντ. Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε μια αξιολόγηση του καθεστώτος ως ίσχυε μέχρι τώρα. Πρέπει να δούμε τι μας συμφέρει εμάς καταρχήν. Και γνωρίζω τι φρονούν οι Ρώσοι επιχειρηματίες που είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα δεν νομίζω ότι μια απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για αυτούς θα ήταν συμφέρον μας. Πρέπει πρώτα να ζητήσουμε από την Κομισιόν να δει τα πρώτα χρόνια των διευκολύνσεων των θεωρήσεων τι απέδωσαν. Με εντυπωσίασαν αυτά οι εντυπώσεις του Βέρνερ Σούλτς γιατί είχαμε πάει μαζί στη Ρωσία. Ας μην επαναλάβω αυτά που είπε, απλώς συμφωνώ για τις θεωρήσεις, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε αν θα ισχύει για το σύνολο της ρωσικής επικράτειας η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Θα ήταν πολύ άσκημο να κάνουμε αυτό που κάναμε και στην Απχαζία και ως αιτία όπου δώσαμε καθεστώς ελευθέρωσης βυζών, αλλά όχι στη Γεωργία. Πρέπει και αυτό να το δούμε. Ο Χάνες μας είπε ότι η έκθεση δεν είναι τόσο θετική όσο θα έπρεπε, όσο θα ήθελε. Ναι, ναι, βγαίνει, τελειώνω, τελειώνω, την πρόταση να τελειώνω. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να μην έχουμε δύο μέτρα αλλά και δύο σταθμά. Πρέπει τη Ρωσία να τη δούμε με τα ίδια κριτήρια με τα οποία βλέπουμε τη Γεωργία, του Αζερμπαϊτζάν γιατί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χειροτερεύει στη Ρωσία και η μόνη ελπίδα είναι το δημοκρατικό κίνημα ή τα δημοκρατικά κινήματα να ενδυναμωθούν. Να, αυτά μπορούσα να σας πω σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σφόμποντα, ο οποίος έχει θέσει στερεές βάση για ένα ψήφισμα. Όπως είπατε, ο χαρακτήρας της εταιρικής μας σχέσης είναι ακόμα ανοιχτός. Οι προϋποθέσεις για μια στρατηγική εταιρική σχέση δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του ψηφίσματός μας. Όπως ελέγχθη υπάρχουν ακόμα κάποια ψήγματα ε, συμπεριφοράς ψυχρού πολέμου στις σχέσεις μας. Για μένα ένα σημαντικό ερώτημα είναι το κεφάλαιο Β από την ε, πρώτη σελίδα όπου αναφέρουμε ότι, είναι, υπάρχει αλληλεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά. Για το πολιτικό τομέα εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα σίγουρος γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πολιτικά μας συστήματα. Θα μπορούσε να το κατανοήσει με διαφορετικό τρόπο το πολιτικά. Αλληλένδετα τα δύο μέρη. Ίσως είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιήσει κανείς καθόλου αυτό τον όρο, το πολιτικό. Μια δεύτερη ιδέα είναι ότι πρέπει να είμαστε ίσως πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το τι εννοούμε εξυγχρονισμό. Είναι σαν να μιλάμε για την περιστρόικα πριν από 25 χρόνια που ήταν μια έκφραση που προέκυψε από μια πλήρη οικονομική και κοινωνική κρίση στη Ρωσία. Η έννοια του εξυγχρονισμού είναι μια πολύ αμφίσιμη και ασαφής έννοια. Αν χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια διατύπωση θα πρέπει να την συνοδεύσουμε με περισσότερη ουσία. Πώς λοιπόν θέλουμε να κατανοήσουμε την έννοια του εξυγχρονισμού. Εγώ ε, χαίρομαι για το γεγονός ότι αναφέρονται σε αυτό το σχέδιο ορισμένα στοιχεία ερεσιμότητος. Αυτό πρέπει να είναι και η βάση της εργασίας μας, ώστε να είμαστε ρεαλιστές και επικοδομητικοί στις σχέσεις μας. Παραδείγματος χάρη για την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ θα είναι αυτό μία από τις προϋποθέσεις. Επίσης ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για την ενέργεια, διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια συμφωνία, ιδίω μια ρήτρα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρόποι να βαθμονομείται αυτή η προστασία με benchmarks. Θέλω επίσης να προσθέσω και δύο ιδέες. Καταρχήν, για τις συνθήκες της λειτουργίας των δυτικών εταιριών στη Ρωσία και των επενδύσεων, για την διαφάνεια και την αμοιβαιότητα, γιατί αυτό συνδέεται άμεσα με το θέμα της διαφθοράς. Πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι ότι οι δυτικές εταιρείε θα πρέπει να προσαρμοστούν στη ρωσική κατάσταση και να συμμετάσχουν σε διεφθαρμένες συναλλαγές. Το δεύτερο θέμα το οποίο με απασχολεί είναι ότι ζητάμε τη Ρωσία να σεβαστεί τα δικαιώματα των ε, γειτόνων της για ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε για τη Ρωσία που υπάρχει μια ισχυρή παρουσία και επιρροή της Ρωσίας στις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γεωργία. Και ένα πρόσθετο στοιχείο θα πρέπει να είναι να κατανοήσουμε ότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους σχεδόν τους τομείς να σεβαστεί την συμφωνία του Αυγούστου 2008 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για το πέρας των εχθροπραξιών στη Γεωργία. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να πάνε ακόμα στις υποαπόσχηση περιοχές. Αυτό είναι μια ταπείνωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. που δεν παρέχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Σφόμποντα. Νομίζω ότι η δική του χώρα καταγωγής ήταν πραγματικά ένα παράδειγμα χώρας από την οποία η Ρωσία έπαιρνε δυνάμεις. Κάποτε ο Μπερλοσκόνη είχε μιλήσει ότι θα πρέπει σε κάποια φάση η Ρωσία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένας Ρώσος πολιτικός είπε ότι η Ρωσία δεν θα μπει σε άλλον τις ενώσεις, αλλά φτιάχνει τις δικές της ενώσεις. Και νομίζω ότι βλέπω τι προσπαθεί να κάνει τώρα να ε, συγκολήσει τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, την Ουκρανία εγώ πάντα θαύμαζα το λαό της Ρωσίας, τον πολιτισμό της Ρωσίας και η Ρωσία είναι στρατηγικός εταίρος όπως και η Κίνα επί τη βάση κοινών οικονομικών και ε, συμφερόντων και συμφερόντων ασφαλείας. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τη Συρία, με το Ιράν, με τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Προσπαθεί να συνεργαστεί η Ρωσία και με τη νέα Σερβία του Προέδρου Νίκολιτς και όλα αυτά γίνονται και μέσω της χρήσης του φυσικού αερίου. Υπάρχουν και άλλα μέρη όμως ε, στο Νότιο Κάφκασο όπου είμαστε ανταγωνιστικοί με τη Ρωσία και θεωρώ ότι τελικά η Ρωσία έχει μια αμφιλεγόμενη τάση θα έλεγα να σέβεται με το δικό της τρόπο την δημοκρατία η συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΝΟΑΣΑ νομίζω ότι ε, είναι οριακές σε σχέση με το σεβασμό του κανονισμού λειτουργίας τους. Δεν έχω ψευδεστήσεις λοιπόν ότι η Ρωσία βλέπει τον κόσμο με ένα σοβιετικό κατά κάποιο τρόπο με μια σοβιετική μέθοδο και αγνοεί τελικά τις βασικές αξίες που μπορεί να μοιράζεται ή να μην μοιράζεται με τη Δύση. Οπότε τι γίνεται με τη Ρωσία και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κοιτάμε να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι σε κάθε χώρα όταν μιλάμε βλέπουμε ότι τα θέματα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της, ε, του κράτους δικαίου κτλ. είναι στην ουσία κάτι το πάρα πολύ επιφανειακό, είναι ένα φιλοσικής. Και το ίδιο πιστεύουν και οι Ρώσοι. Δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ότι η Ρωσία θα σεβαστεί γενικά τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά οι Ρώσοι μας χρειάζονται όπως και εμείς τους χρειαζόμαστε σε πάρα πολλά διεθνή ε, θέατρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι παρατηρήσεις του κυρίου Σβόμπο uh, uh, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν πιστεύουμε στην πρόοδο και στην αποστολή μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Δεν μπορούμε εμείς να υπογραμμίσουμε όπως είπε ο κύριος Σβόμποντα τη στρατηγική σχέση που πρέπει να έχουμε με τον συγκεκριμένο εταίρο. Να μην το θεωρούμε αυτό μια αναγκαιότητα de facto χωρίς να μοιραζόμαστε τίποτα άλλο με τη χώρα αυτή βλέπουμε ότι η χώρα αυτή λειτουργεί σαν μια χώρα η οποία προσπαθεί να κάνει τον κόσμο χειρότερο. Βλέπουμε ότι καταλαμβάνει στρατιωτικά γειτονικά εδάφη και δεν βοηθά στην προσπάθεια να καταστήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο καλύτερο. Ας θέσω λοιπόν και κάποια άλλα σημεία στην αιτιολογική σκέψη α του κυρίου Σβόμποντα για την εταιρική μας στρατηγική σχέση θα ήθελα να πω ότι εδώ μιλάμε για μια ευχή. Θα θέλαμε να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική σχέση σε θεμελιώδη θέματα. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμεθα, αλλά Τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για προώθηση της στρατηγικής σχέσης. Να πω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε ε, κάθε δυνατότητα εταιρικής σχέσης όπου σημειώνεται πρόοδος, όχι εκεί όπου υπάρχει το αντίθετο. και σαν παράδειγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εταιρική σχέση με τη Ρωσία στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η διεθνή ειρήνη λοιπόν θα πρέπει να είναι κανονικά ο κοινός στόχος μας με τη Ρωσία, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να δείξουμε στο έγγραφο αυτό και το οποίο δεν διαφαίνεται είναι το θέμα της εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας να επανέλθουμε στις θέσεις τις οποίες είχαμε το 2008. Ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αμφισβητείται από την αριστερά μας σήμερα βέβαια, σχετικά με τη θέση της Ρωσίας και τα κατεχόμενα εδάφη. Το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει και δεν μπορούμε να το κρύβουμε. Τώρα για τις σωστούς κανόνες λειτουργίας του πιστοτικού συστήματος και των εμπορικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η οικονομική συνεργασία σαν πολιτικό όπλο. Όλα αυτά είναι το στους οποίους μένει να υπάρξει πρόοδος. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Σφόμποντα για την ε, ιδιαίτερα καλά προετοιμασμένη πρότασή του. Εγώ έχω κάποιο βαθμό αισιοδοξία. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει με τους Ρώσους συναδέλφους μας ότι δεν μας ενδιαφέρει μοναχά το θέμα της τεχνικής προόδου και του εξυγχρονισμού, αλλά και για τον εξυγχρονισμό της σύνολης ρωσικής κοινωνίας. Έχω λοιπόν κάθε ελπίδα ότι μπορούμε να επιτύχουμε πραγματικά μια συνεννόηση σε στρατηγικό επίπεδο. Έχουμε βέβαια σε πολλά σημεία διαφορές σε στρατηγικά σημεία και απόψεις. Είδα αυτή την νομοθεσία που αφορά τις ΜΚΟ και τους ξένους πράκτορες μέσα εισαγωγικά, το νόμο αυτό που περνάει από την Τούμα. Αλλά αυτός ο νόμος είναι τελείως διαφορετικός από την δική μας αντιμετώπιση του πώς πρέπει να λειτουργήσει μια ελεύθερη κοινωνία. Αν το κείμενο αυτό παραμείνει με αυτή τη μορφή, αν αυτός ο νόμος τεθεί σε εφαρμογή, αυτό θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω πόλωση της ε, ρωσικής κοινωνίας. Θα έχουμε λοιπόν άτομα τα οποία θα πρέπει να καταγράφονται στα Μητρώα ως ξένοι πράκτορες μέσα εισαγωγικά και αν δεν το κάνουν αυτό, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν κυρώσεις. Επομένως, εγώ πρέπει να συμφωνήσω και με την κυρία Όμεν Ρόιτεν ότι αυτό το ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι σύντομη και στεναρή. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα κατάλογο με θέματα τα οποία είναι δευτερεύοντα. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικά, στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα βάσει των οποίων μπορούμε να οικοδομήσουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση και όχι να λέμε ότι δεν μπορούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική σχέση για θέματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου και θα ήθελα της ε, διεύθυνσής μου και θέλω να σας πω ποια είναι η θέση μας. Εμείς ζητάμε την επίτευξη μιας ε, καινούργιας συμφωνίας με ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο όμως όπου δεν έχει σημειωθεί πρόοδο στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τις επενδύσεις και για τα ενεργειακά βέβαια. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κεφάλαιο αν θέλουμε όντως να υπάρξει μια πραγματικά νέα συμφωνία που να καλύπτει όλες τις πτυχές των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Κατά τις συζητήσεις μας με αυτούς σημειώσαμε ότι το πρώτο βήμα προς τα εμπρός ήταν η έγκριση σήμερα από την Δούμα του γενικότερου πλαισίου. Πρέπει όμως να το ξεπεράσουμε αυτό για την ένταξη της Ρωσίας στον ΟΕ. Έχουν υποθεί πολλά για την Τελωνιακή Ένωση και δεν μπορούν να μετακινηθούν πολύ περισσότερο από τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία για να δούμε τι θα γίνει. Και είπαμε στους Ρώσους συνομιλητές μας σε ανώτατο επίπεδο ότι η εντολή μας είναι για συμφωνία με τη Ρωσία, όχι για μια απλή ακυταλωνιακή ένωση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, πώς θα τελειώσει η διαπραγμάτευση. Η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι που το συζητήσαμε και σήμερα εδώ μέσα σε μια ρωσική, με μια ρωσική ομάδα αντιπροσωπεία η σημασία της κοινωνίας των πολιτών μειώνεται λόγω νομοθετημάτων που έχουν εγκριθεί πρόσφατα και που προτίθενται να περάσουν οι Ρώσοι και που τα γνωρίζουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και η Πάτη εκπρόσωπος εξέφρασε τις ανησυχίες της αυτές για και μιλήσαμε, συνομιλήσαμε και με τους εκπροσώπους της Δούμας και της κυβέρνησης για τα προβλήματα που βλέπουμε να υπάρχουν αν εφαρμοστούν τέτοια νομοσχέδια. Να αυτά, αυτά. Θέλω να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σφόμποντα. Για να είμαι σύντομος λέει ο κύριος Σφόμποντα. Νομίζω ότι είναι σαφής η θέση μου. Έχουμε μια συμφωνία που ισχύει ήδη. Αν θέλουμε να κάνουμε μια νέα συμφωνία με την ε, Ρωσία, αυτό θα πρέπει να έχει μια προσθέμενη αξία. Δεν πιστεύω ότι πρέπει κάτω από οποιοδήποτε συνθήκε να έχουμε μια νέα συμφωνία, αν δεν έχει προσθέμενη αξία. Δεύτερον, είπα σαφώ ότι αυτή τη στιγμή δεν χωρούν οι προϋποθέσεις μιας στρατηγικής ε, ε εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Δεν πρέπει να ο κύριο Στανσπέργκη. Θέλουμε να έχουμε μια τέτοια στρατηγική σχέση, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εκπληρωθούν για να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η έννοια της ε, σχέσης σύνδεσης ήταν ένα σφάλμα. Όπως είπε και η κυρία Όμεν Ρόιτεν, δεν είναι αυτό το οποίο επιζητούμε εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία και κάποια πρόοδος στη Ρωσία. Δεν έχω την ίδια ε, θέση με τον κύριο Σούλτς ότι είναι όλα αρνητικά. Επίσης, στην έκθεση, στην σχέση για τελωνιακή ένωση διαπραγματευόμαστε με τη Ρωσία όχι μια ευρύτερη τελωνιακή ένωση που περιλαμβάνει τη Ρωσία. Στα σημεία αυτά που ανέφερε ο κύριος Σούλτς για τα θέματα των προξενικών θεωρήσεων, όπως και στην περίπτωση της ε, Γεωργίας και της Ουκρανίας και με τη Ρωσία έχουμε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ταχαίως σε μια λύση και με τη Ρωσία. Τα θέματα της πολιτικής αλληλεξάρτησης συμφωνώ ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είχαμε μια, σαφή, να είχαμε μια σαφέστερη διατύπωση έχουμε μια οικονομική αλληλεξάρτηση και θα έπρεπε να υπάρχει και μια μεγαλύτερη πολιτική αλληλεξάρτηση, αλλά αυτό δεν ισχύει. Σήμερα θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε καλύτερα για το θέμα του εξυγχρονισμού. Επίσης, δεν είναι μονάχα μια οικονομική ε, υπόθεση ο εξυγχρονισμός, αλλά είναι και ένα πολιτικό ζήτημα. Χρειάζεται ίσως εδώ μια καλύτερη διατύπωση και επίσης το σημείο το ότι η Ρωσία πρέπει να αφήσει τους γείτονές της να λειτουργήσουν αυτόνομα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ε, αυτονόητο. Θέλουμε να έχουμε συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει και την αυτονομία των, των ε, όμορων της χώρων και να μην, τις να μην τις επηρεάζει. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ισχυώδεις συζητητές για αυτή τη συζήτηση και να πω επίσης ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα των ΜΚΟ, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επομένως θα πρέπει να επιμείνουμε στα σημεία αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει δεν θέλω να μιλήσω τώρα για θέματα όπως οι παιδείς και τα λοιπά. Αν δεν υπάρξει πρόοδος σε όλα αυτά τα στοιχεία, καμία συμφωνία δεν θα μπορεί να είναι αποδεκτή για το κοινοβούλιο μας. Και επομένως για αυτό το λόγο δεν πρέπει εμείς να κάνουμε ένα κατάλογο ονείων που να περιλαμβάνουμε όλες τις δυνατές πτυχές. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, θα πρέπει να ξέρουν οι διαπραγματευτές ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το Κοινοβούλιο θα δεχτεί μία συμφωνία. Δεν θέλουμε να απορρίψουμε εκ των υστέρων μία ε, συμφωνία με τη Ρωσία. Πρέπει να πούμε εκ των προτέρων στους διαπραγματευτές ότι κοιτάξτε δείτε εδώ πέρα έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την θετική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ο μηχανισμό με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Όχι να πούμε μόνο ότι έχουμε μία σύσταση ή μία άποψη, αλλά ότι έχουμε σαφεί προποθέσει τι οποίε θεσπίζουμε ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει μία συμφωνία με τη Ρωσία και θα ήταν λοιπόν σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν θέλουμε μια συμφωνία παστησία και ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. Αυτά λοιπόν, εγώ περιμένω τις τροπολογίες σας και ευχαριστώ όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος ε, Μπροκ, χωρίς μικρόφωνο βέβαια. Τροπολογίες μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου καταληκτική τροπολογία. Μπορείτε με κάθε ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσετε το καλοκαίρι σας για να σκεφτείτε για αυτές και θα ψηφίσουμε στις 11 Οκτωβρίου. Σημείο 22, ευχαριστώ τον κύριο Σόμποντα προηγουμένως. Ερχόμαστε στην υπόθεση Μαγνίτσκι. Η κυρία Όγιουλαντ θα λάβει το λόγο για παρουσιάσει το θέμα αυτό. Όλοι γνωρίζουμε τα θέματα αυτά, έχουμε μιλήσει πολύ για τη Ρωσία και θα συνεχίσω προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το έγγραφο αυτό με ευρύτητα πνεύματος. δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια επιθετική στάση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, αλλά είναι κάτι που πρέπει να μεταφέρει σημαντικά μηνύματα προς τους Ρώσου εταίρου ότι δεν θέλουμε εμείς να υπάρχει έκπληνση χρημάτων σε εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλουμε ε, τα βρώμικα αυτά χρήματα να επενδύονται σε αγορές. Δεν θέλουμε να έχουμε σχέσεις με αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σκοτώνουν τους Ρώσους δικαστές, δεν θέλουμε να έρθουν στη, στα ευρωπαϊκές χώρες μας. Να υπενθυμίσω ότι το 2010 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της ετήσιας έκθεσης, ήδη από τότε είχαμε τον λεγόμενο κατάλογο Μαγνίτσκι που αποτελείται από 50 θα έλεγα ανθρώπους οι οποίοι είχαν ε, σκοτωθεί ενώ βρισκόντουσαν υπό προσωρινή κράτηση. Και είχαμε ζητήσει από το Συμβούλιο να επιβάλλει εις βάρος αυτών των 60 α, τις απαιτούμενες κυρώσεις. Εν τω μεταξύ όμως, Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι η διαφθορά στην Ρωσική Ομοσπονδία έχει αυξηθεί, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν και αυτές αυξηθεί. Υπήρξαν διώξεις εις βάρος της μητέρας και της οικογένειας του Μαγνίτσκι. Νομίζω εν πάση περιπτώσει ότι καιρός είναι να θέσουμε το θέμα εκ νέου και να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, σε επίπεδο θεωρήσεων εις βάρος αυτών οι οποίοι ήταν ένοχοι και στον θάνατο τον δικό του. Αντίθετα δεν τιμωρήθηκαν αλλά πήραν προαγωγή πήραν μετάλλια. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε κάποια μορφή κυρώσεων εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Επίσης και κυρώσεις σε επίπεδο οικονομικών αγαθών που μπορεί να έχουν στις χώρες της mm. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι επί τη βάση ανεξαρτήτων πληροφοριών, έγκυρων πληροφοριών, να πάρουμε περιοριστικά μέτρα και εις όλους όλων αυτών των Ρώσων οι οποίοι συμμετέχουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να φροντέξουμε είναι το ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει ήδη περάσει τον νόμο τον λεγόμενο Μαγνίτσκι και τώρα προχωρούν, έχει, θα φτάσει στην Ολομέλεια ε, για να υπάρξουν και τροπολογίες στον λεγόμενο νόμο Μαγνίτσκι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και σε σχέση με το πάγωμα ας πούμε ποσών που μπορεί καταθέσεων που μπορεί να έχουν υψηλά ιστάμενοι Ρώσοι εξωματούχοι σε Αμερικανικές τράπεζες ε, αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς ε, και στις τράπεζες ε, θηγατρικές ή που ανήκουν στην ίδια εταιρεία εν πάση περιπτώσει και λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν δύο εβδομάδες ήμουνα στη Ουάσιγκτον και οι συνάδελφοι στη Γερουσία και από τα δύο κόμματα και από πλευράς δημοκρατών και από πλευράς των συντηρητικών πήραν μέρος στη συζήτηση. Η συζήτηση ήταν πληρεστάτη. Μιλήσαμε για την εταιρική σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, για τις κοινέ αξίες και τις κοινέ ανησυχίες της ε, διατλαντικής αυτής συμφωνίας. Πρέπει να τηρήσουμε και να έχουμε κοινέ θέσεις απέναντι στους Ρώσους και φυσικά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους Ρώσους. Λοιπόν, περιμένω να προχωρήσει η συζήτηση στο συγκεκριμένο σημείο. Θα το συζητήσουμε για να το υιοθετήσουμε τον Σεπτέμβριο σε μία από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, ο πρόεδρος. Θα είμαι πολύ σύντομος, λέει ο κύριος ε, ε, Σαλαφράνκα, ο κύριος πορτασέβιτς, ο οποίος ως κοιόδης εισηγητής για το θέμα αυτό, μου ζήτησε να μεταφέρω την ε, γνωμοδότησή του, υποστηρίζει αυτή την γνωμοδότηση και εμείς θέλουμε να πούμε στην συγγήτρια ότι συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότηση το οποίο συζητούμε, στο σχέδιο έκθεση μάλλον, θα ήταν όμω ενδιαφέρον να σκεφτούμε και για μερικέ συμπληρωματικέ μνήε. Στην παράγραφο 1 θα ήταν θετικό να πούμε πέραν του γεγονότος ότι είναι μια τραγική περίπτωση να, και ότι πρέπει να έρθουν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη να ζητήσουμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τροποποιήσουν το δικαστικό του σύστημα. Και μου λέει επίσης ο κ. Προτασίεβιτς ότι έχει κάποιες ε, αμφιβολίες για την τελευταία φράση της παραγράφου 2 που λέει και άλλα περιοριστικά μέτρα και θα στείλει στην ε, εισηγήτρια ορισμένα πρόσθετα σχόλια για το θέμα αυτό. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό μετά από τη συζήτηση που προσπαθούμε να έχουμε για τις σχέσεις με τη Ρωσία θα ήταν να καταλήξουμε σε κάποια μορφή ερεσιμότητος σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Να υπάρξει λοιπόν αυτή η σύνδεση από τον ε, εισηγητή, τον κύριο Σφόμποτα, μου φαίνεται ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να, να γίνει και σε αυτή την περίπτωση, στην έκθεση της κυρίας Όγιουλαντ. Νομίζω λοιπόν ότι μια λογική κατάληξη αυτής της, προ... της σύστασης προς το Συμβούλιο ίσως θα ήταν πιο λογικό να βάλουμε το δεύτερο σημείο πριν από το πρώτο σημείο, να αναστρέψουμε τη σειρά. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και θέλω να σας μεταφέρω αυτά τα οποία λέει ο κύριος ε, Προτάσιβης και να σας τονίσω ότι η ομάδα μου συμμερίζεται τις απόψεις που τις Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Όγιουλαντ για την πλήρη αυτή παρουσίαση για την περίπτωση Μαγνίτσκι. Υπάρχει φυσικά και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει ότι πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εμπλεκομένων αξιωματούχων. Υπάρχουν όμως κάποια ε, εθνικά κοινοβούλια τα οποία έχουν ακολουθήσουν τους Αμερικανούς και έχουν επιβάλει τέτοιες μορφές ε, απαγορεύσεων ταξίδιων ορισμένων αξιωματούχων. Δεν είναι, δεν είναι κάποια μεμονωμένη περίπτωση, είναι απλώς μια ακραία περίπτωση για την ε, αντιμετώπιση των ατόμων που μάχονται κατά της διαφθοράς στη Ρωσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει μια μέθοδος ώστε, όπως παραδείγματος χάρη έγινε και την περίπτωση του Αλεξάνδρ Λέμπεντεφ, ο οποίος αγωνίστηκε κατά της διαφθοράς, και στην περίπτωση του κυρίου Ζόκολοφ, του αρχιστάκτη της Νόβα Γιαγκαζέτα, όπως σας είπα, τον απαγάγαν, τον πήγανε σε ένα δάσος και τον συνάντησε εκεί ο Γενικός Εισαγγελέας Ρωσίας και τον ε, απείλησε με εκτέλεση. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα σας φαίνονται απίστευτα και απίθανα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στη Ρωσία. Αυτά λοιπόν κάνουν την περίπτωση Μαγνίτσκι μια ε, ιδιαίτερα τραγική περίπτωση, τον εκτελέσαν στη φυλακή, αλλά και πάλι δεν πρέπει να το δούμε σαν ένα μεμονωμένο γεγονός. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μέτρα και θα πρέπει να επιμείνει να υπάρξει έρευνα για το θέμα αυτό. Η απαγόρευση λοιπόν για τα ταξίδια αξιωματούχων που είναι εμπεπλεγμένοι σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η Ρωσία απλώς έχει επενέσει μετά θάνατον τη δράση του Μαγνήσικη. Αυτό δείχνει το πόσο καυκικά και παράξενα είναι τα πράγματα που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ τον εισαγητή για την πρωτοβουλία του που είναι πολύ επίκαιρη Ήταν καιρός να κάνουμε κάτι επιτέλους. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ο αριθμός παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αυξηθεί πολύ, καθώς και η διαφουθορά. Πρέπει να αρχίσουμε με την περίπτωση Μαγνίτκη, γιατί είναι η πιο καλά τεκμηριωμένη, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες. Αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε πολιτικά και που θα μπορούσε να αποβεί ωφέλιμο να αλλάξει τη συμπεριφορά της ρωσικής διοίκησης ώστε να μεταρρυθμίσει το δικαστικό της σύστημα για περισσότερη διαφάνεια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει κάτι. Γι' αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε από αυτού το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, τότε θα είχαμε πολύ περισσότερο κύρος. Ευχαριστώ. Uh, thank you, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ σέβομαι ιδιαίτερα την κυρία Όγιολαντ για την πρωτοβουλία αυτή. Στην αρχή δεν ήμουν βέβαιος αν χρειαζόταν κάτι τέτοιο ή αν θα ήταν αποτελεσματικό, αλλά πίστηκα. Βέβαια είναι άγνωστο, άγνωστα τέτοια πράγματα. Εδώ ούτε είναι ακριβώς δικαιοδοσία του Κοινοβουλίου, γιατί πρόκειται για τρίτες χώρες, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να δούμε αν περάσει το μήνυμα στη Ρωσία ίσως και σε άλλες χώρες ότι τα παίρνουμε σοβαρά όσα λέμε για στήριξη των θεμελιωδών παλιτικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ρωσία που υπόθηκε επανειλημμένος ότι είναι και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Φανταζόμουν ότι οι οργανισμοί αυτοί κάτι κάνανε για να γίνει σεβαστή η νομοθεσία που ισχύει στις ίδιες αυτές τις χώρες, αλλά φαίνεται ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και τελικά η διεθνής καμπάνια που έγινε για την περίπτωση Μαγνίτκι μας δίνει την ευκαιρία να πούμε και εμείς κάτι γι' αυτό. Και στη Βουλή των Κοινοτήτων θα προταθεί κάτι ανάλογο, όχι δεσμευτικό βέβαια. Και η Βρετανική κυβέρνηση, αν και είπε ότι δεν θα το δεχτεί επισήμως, θα αναγκαστεί να λάβει υπόψη της όλους όσους συνυπογράφουν Ως πολιτική χειρονομία λοιπόν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και ελπίζω να υποστηριχθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες στην Ολομέλεια γιατί αλλιώς θα χάσει την πολιτική, το πολιτικό του νόημα. Ελπίζω λοιπόν να υποστηριχθεί από όλο το κοινοβούλιο. Και το Κρεμλίνο αυτή τη φορά αντί να γνωρίσει τα πράγματα θα αναγκαστεί να προσέξει τι λέμε. Όταν ήταν πρόεδρος ο Μετβέντεφ είχαν ακουστεί υποσχέσεις ότι θα αναθεωρηθεί ή θα εξεταστεί η υπόθεση Μαγνίτσκι αλλά Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα ούτε αποδόθηκε δικαιοσύνη στα μέλη της οικογένειας του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από τη δική μας πλευρά θέλουμε να τονίσουμε ότι και εμείς είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη προόδου για την έρευνα της περιπτώσεως Μαγνίτσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πάντα επιτάπητο στο ζήτημα αυτό ακόμα και σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Ο πρόεδρος Φαν Ρομπόη έστειλε μια επιστολή πριν από την τελευταία διάσκεψη κορυφής με τη Ρωσία για να τονίσει το πρόβλημα αυτό και είπε πολύ σαφώς ότι αυτή η περίπτωση είναι εμβληματική της κατάστασης του κράτους δικαίου και της δικαστικής εξουσίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και παρότρινε τον Ρώσο Πρόεδρο να συνεχίσει και να περατώσει τις έρευνες και έθεσε επίσης και το θέμα της ε, μεταθανάτιες έρευνας για τον κύριο Ματσκνίσκη και της ε, σύλληψης οικογένειάς του. Εμείς λοιπόν θέλουμε να παροτρύνουμε τη Ρωσία να προχωρήσει σε αυτή την έρευνα και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τους ενόχους. Η επόμενη ευκαιρία θα είναι η συνάντηση με την Ρωσική Ομοσπονδία που θα γίνει σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Για το θέμα των κυρώσεων είναι φυσικά μια τελική καταφυγή, ultima ράσιο σε διεθνείς σχέσεις και θα πρέπει οι κυρώσεις αυτές να ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήρες γραμμές που έχουμε υιοθετήσει για κυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τις προθεσμίες για τις τροπολογίες μέχρι τις 29 Αυγούστου. 20 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλα τρία σημεία της σημερινής διάταξης. Μετά από συζήτηση με τον εισηγητή, θα ήθελα να έχουμε μια πολύ σύντομη συμφωνία για την ε, εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και το Περού και για το θέμα της Κεντρικής Αμερικής και θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να συζητήσουμε με τον πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλγερία. Κύριε Σαλαφράγκα, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μπορέσουμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε αυτό το θέμα και θα ήθελα εγώ να θέσω δύο ζητήματα σε μια κοινή συζήτηση γιατί εγγράφονται στην ίδια προβληματική και έχουμε τον ίδιο στόχο παρά το γεγονός ότι ένα από τα θέματα αυτά εγγράφεται μέσα στον κατάλογο των αρμοδιοτήτων της δικής μας Επιτροπής γιατί έχει την φύση μια συμφωνίας σύνδεσης και το άλλο είναι μια συμφωνία η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και εμεί είμαστε απλώ γνωμοδοτική επιτροπή. Είναι απαραίτητο να εγγράψουμε λοιπόν και τι δύο αυτέ πτυχέ, τα δύο θέματα σε μια ιστορική πορεία για, την, για τον διάλογο τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική και τη ομάδα του Ρίο και επίση του μηχανισμού του εμπορικού που διέπουν τα θέματα αυτά. Βρισκόμαστε στην τέταρτη γενιά συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών τη Λατινική Αμερική. Ξεκίνησαμε με τη συνεργασία και τη βοήθεια για την ανάπτυξη. Το δεύτερο περιλαμβάνει τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία επίση. Η τρίτη γενιά είχε και τη δημοκρατική ρήτρα που αποτελέσε ένα σημαντικό στοιχείο των συμφωνιών που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι τρίτε χώρε. Η τέταρτη τώρα γενιά διατηρεί τη δημοκρατική ρήτρα, αλλά εστιάζει περισσότερο στην βαθμία φιλελευθερωποίηση των συναλλαγών. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω απλώ κύριε Πρόεδρε ότι αυτέ οι συμφωνίε θέλουν να ξεπεράσουν ένα καθεστώς μονομερών παραχωρήσεων που ξεκίνησε από τα μέτρα τα οποία δόθηκαν τα ευνοϊκά μέτρα προς την Κολομβία και άλλες χώρες όπως το Περού στον αγώνα κατά του εμπορίου, της εμπορίας ναρκωτικών και θέλουν να δώσουν μια προτιμησιακή πρόσβαση στα προϊόντα των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές με ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο ε, καθεστώς το οποίο ξεπερνάει το προηγούμενο απόλυτα μονομερές καθεστώς, το οποίο είχε πολλά αστάθμητα στοιχεία. Επίσης, οι συμφωνίες αυτές, αυτό το οποίο επιζητούν, είναι να τοποθετήσουν τις σχέσεις μας με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και την Κολοβία και το Περού σε ένα πιο όριμο πλαίσιο τη στιγμή που οι χώρες αυτές προχωρούν περισσότερο προς αμοιβαίου χαρακτήρα συμφωνίες. Όπως ξέρουν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, οι διαπραγματεύσεις αυτές για την επίτευξη αυτών των συμφωνίων έχουν φτάσει στο τέλος και έχουν μονογραφηθεί το Μάιο του 2010 και εκτότε έχουν περάσει δύο έτη χωρίς το Κοινοβούλιο μας να κληθεί ακόμα να εκφέρει γνώμη για τα θέματα αυτά. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιο προβληματισμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την ανεπάρκεια των διαδικασιών μας, όχι του Κοινοβουλίου, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να εκφέρουμε την απόψή μα. Αυτή είναι φυσικά η άποψη του εισηγητή. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ποιε είναι οι διαδικασίες όταν πρέπει να υπάρχει συμφωνία σύμφωνης γνώμης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από αυτά τα οποία διαπραγματεύεται η Κομισιόν εξ ονόματο των 27 κατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να πούμε κάτι μέσω των ψηφισμάτων μας, μέσα στο πλαίσιο αυτό. Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω με τους σκιώδεις εισηγητές των διαφορών πολιτικών ομάδων το πώς θα μπορούσε να διατυπωθεί αυτό το ψήφισμά μας. Και ως εισηγητής επίσης γνωμοδότησης για τη συμφωνία με το Περού και την Κολομβία, θεωρώ ότι όπως όλοι έχουν καταλάβει θα είναι θετική η γνωμοδότησή μου. Οι συμφωνίες αυτές ξεπερνούν τις προηγούμενες ασυμμετρικές συμφωνίες, δημιουργούν ένα καλύτερο πλαίσιο και βελτιώνουν και την πρόσβαση για την λατινοαμερικανική πλευρά θα είναι εξάλλου σημαντική και θετική για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό τονίζω ότι εγώ είμαι υπέρ τη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτέ τι συμφωνίε και είμαι πάντα έτοιμο να συνεργαστώ με τα άλλα πολιτικά κόμματα για την διατύπωση ενό ψηφίσματο το οποίο θα καλύπτει όλε τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να λάβω το λόγο εξ ονόματο του Ραϊμόν Οβιόλς από τη Σοσιαλιστική Ομάδα που δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα το απόγευμα και τον εκπροσωπώ σήμερα. Κάποια θέματα διαδικασίας. Νομίζω ότι υπήρξε κάποια σύγχυση στην διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την ε, έκθεση, γιατί ήταν η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων η οποία πρότεινε ένα ψήφισμα και όχι μια προσωρινή έκθεση όπως αποφάσισε η συνέλευση των Προέδρων. Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις και ένα πλαίσιο για την διεθνή αυτή συμφωνία. Επίσης υπήρξε κάποια σύγχροση αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου για τις συμφωνίες αυτές με την Κολοβία, το Περού και την Κεντρική Αμερική. Και το ψήφισμά μας θα πρέπει να είναι ένα ψήφισμα από την Επιτροπή Εξωτερικών, η οποία έχει μια ιδιαίτερη ε, ευαισθησία στο να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. Και επί της ουσίας τώρα έρχομαι. Ο κύριος Ομπιόλ θέλει να συγχαρεί τον εισηγητή για το σχέδιο ψηφίσματός του που είναι μια πολύ καλή βάση για να επιτύχουμε τους στόχους μια σχέση σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής. Είναι η πρώτη συμφωνία η οποία είναι διπεριφερειακού χαρακτήρα που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη περιοχή, την Κεντρική Αμερική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, αλλά υπάρχει ένα κεφάλαιο για πολιτική, τον πολιτικό διάλογο που τονίζει η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωση. Θα ήθελα να έχω την ίδια ευκαμψία σε σχέση με τον χρόνο όπως είχαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Είπαμε να το κάνουμε αυτό όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ένα λεπτό ίσως. Άντε 30 δευτερόλεπτα παρα, παρα, περισσότερο παρακαλώ. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία επιζητεί σημαντικού στόχου όπω είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση και η κοινωνική συνοχή, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Επίση, ο κ. Σομπιόλ θέτει μια σειρά από τροπολογίε για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία, την αναγνώριση τη ασυμμετρία μεταξύ των δύο αυτών περιοχών είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ιδιαίτερα για τη σοσιαλιστική ομάδα και επίσης για την παρότριση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης τη δυνατότητα να διευρύνουμε στο βαθμό του δυνατό και το, πλαίσιο για το χρονικό πλαίσιο για την ε, κατάσταση τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο και πάλι ο κ. Μπρόκ. Από διαδικαστικής πλευράς πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία, όχι να καθυστερήσει. Εγώ Είχα πάει με μία αντιπροσωπεία των φιλελευθέρων στην Κολομβία πριν από δύο εβδομάδες και μιλήσαμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και τα συμπεράσματά μου όπως και στη σχέδιο γνωματότης του κυρίου Σαλαφράγκα είναι ότι τα πράγματα προχωρούν. Αν δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει βελτίωση. Κατά πολέμηση του εγκλήματος και των ναρκωτικών υπάρχει πρόοδος το Διεθνές Γραφείο Εργασίας επίσης έχει θετική γνωμοδότηση. Βιώσιμη ανάπτυξη υπάρχει. Άρα τελικά πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση του Σαλαφράγκα, να τη φέρουμε στην Ολομέλεια και τελικά καλό θα ήταν να εγκριθεί εκεί. Θα μιλήσω και εγώ στα Ισπανικά. η δική μου ομάδα δεν συμμερίζεται την θετική ανάλυση των άλλων πολιτικών ομάδων και του εισηγητή. Θεωρούμε ότι ακόμα δίνουμε την προτεραιότητα στην ελευθερία του εμπορίου και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρισκόνται σε, δευτερο, σε δευτερεύον επίπεδο. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται και στο Περού και στην Κολομβία. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Κεντρική Αμερική. Δεν μας φαίνεται λοιπόν θετικό και σωστό να προχωρήσουμε με αυτή τη συμφωνία όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να αναφερθώ και σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι μυστικές υπηρεσίες της Κολομβίας, παραδείγματος χάρη, το, το Βέλιο ζητάει μια ερευνητική επιτροπή για τα θέματα αυτά των μυστικών υπηρεσιών της Κολομβίας και για αυτό το θέμα ε, εξετάζεται και από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πιστεύω ότι όσο συνεχίζει αυτή η εξέταση πρέπει να δώσουμε εμεί το καλό έχει σε αυτή τη συμφωνία. Και κάτι ακόμα για την Κεντρική Αμερική. Δεν έχω χρόνο για να μιλήσω για όλα αυτά τα θέματα ενδελεχώ. Στη Συμφωνία τη Κεντρική Αμερική και πάλι προβλέπεται η φιλελευθερωποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό είναι μια βάση που θα ανοίξουμε ουσιαστικά τους ασκούς του αιώλου για να μεταφερθεί και η κρίση και στην χώρα αυτή. Αυτό είναι λοιπόν ένας ακόμα λόγος για τους οποίους η ομάδα μου θα ζητήσει να μην, εγκριθεί αυτή, να μην εγκριθούν αυτές οι συμφωνίες. Θα ήθελα το Σεπτέμβριο όμως να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την γνωμοδότηση που εκπονεί ο συνάδελφος Σαλαφράγκα. I give the floor to Mr. Meyer. Ο κύριος Μάιερ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα για την έκθεσή του. Γνωρίζω, γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η θέση της ομάδας μου, τόσο για τη Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορίου με την Κολομβία και το Περού. Είμαστε εναντίον αυτής της συνθήκης, ιδίως γιατί στην περίπτωση της Κολομβίας και εν μέρη στην περίπτωση του Περού τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικά και το, επίσης γιατί το ελεύθερο εμπόριο όπως ε, διατυπώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες που υπάρχουν, δεν είναι μια ισορροπημένη, συμπληρωματική και δίκαια μορφή εμπορίου που μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις που μαστίζουν αυτές τις χώρες. Εγώ είχα παρουσιάσει στην προηγούμενη έκθεση την έκθεση η οποία οδήγησε στην εντολή διαπραγμάτευσης θεωρώ ότι εγώ αποσύρθηκα τελικά από αυτήν την έκθεση γιατί νομίζω ότι οι προτάσεις μου δεν είχαν ληφθεί υπόψη ιδίως αυτά τα οποία ανέφερα σε σχέση με, την, με το ευαίσθητο της ε, κοινωνίας των κοινωνιών της Λατινικής Αμερικής για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και σε εμπορικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μια ε, ρήτρα η οποία θα ζητά να υπάρχει πληροφόρηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό προβλεπόταν τότε στη δική μου έκθεση, αλλά δεν τηρήθηκε ως το τέλος. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω κύριε Πρόεδρε, εμείς ε, θα καταθέσουμε πάντως τροπολογίες ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν τουλάχιστον κάποια στοιχεία της δικής μας θέσης στο ψήφισμα. Eh, Ο κύριος Μιλανμόν, είναι κάπως ε, παράδοξο να κατηγορείται η Κολομβία για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν και άλλες χώρες βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Και δεν ζητάει κανείς την πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα επιπλέον να τονίσω τη σημασία του να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά οι Ηνωμένε Πολιτείε με τον Ομπάμα και την προστατευτική αυτή στάση που είχαν, παρόλα αυτά δεν είχαν καμιά δυσκολία να κυρώσουν τη συμφωνία ελευθέρων εμπορίου με την Κολοβία. Και σύμφωνα και με τον κύριο Τάνοκ ότι μια χώρα όπως ο Παναμάς που έχει τεράστια σημασία με τη διεύνηση του, του καναλιού του Παναμά θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριο Σαραφράγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την παρέμβασή τους και για τις απόψεις που έχουν διατυπώσει σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις. Επί της ουσίας κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπήρξαν σημαντικέ πρόοδοι σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ δεν πιστεύω όμω ότι πρέπει να έχουμε ένα πατερναλιστικό χαρακτήρα στη στάση μα. Θα πρέπει να βρούμε συμφωνίε οι οποίε συμφωνούν, οι οποίε φέρουν μαζί και το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και των εταίρων μας από την Λατινική Αμερική. Μετά από τις ε, ακροάσεις που κάναμε στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για τα θέματα αυτά, νομίζω ότι έμεινε πάρα πολύ σαφές ότι διάφοροι εκπρόσωποι οι οποίοι ήρθαν και αναφέρομαι στους εκπροσώπους των πολιτών των χωρών αυτών ήταν υπέρμαχοι της σύναψης αυτής της συμφωνίας. Έχει υπογραφεί και από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις λατινοαμερικανικές πλευρές. Καταναβέ ότι υπάρχουν σε ορισμένες πολιτικές ομάδες κάποιες δυσκολίες για να κατανοήσουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν και επίσης και για τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν από μια συμφωνία ελευθερών εμπόριο. Εγώ θέλω να τονίσω περισσότερο τα θετικά στοιχεία και η, η Επιπτώσει που είδαμε στι συμφωνίε με το ελεύθερο εμπορίο με το Μεξικό και τη Χιλή δείχνουν ότι θετικό είναι γενικά το αποτέλεσμα, είναι πιο πολλά τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα τα οποία έρχονται από τέτοιου είδου συμφωνίε. Αυτά λοιπόν είναι η δική μου θέση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάιερ για την ε, επικοδομητική στάση αποχής που είχε σε σχέση με τα θέματα αυτά της, ε, των συμφωνιών. Κατανοώ και τις άλλες αμφιβολίες που διατυπώθηκαν από άλλε πολιτικέ ομάδε για τα ανθρώπινα θέματα, αλλά αυτές είναι πάντα ρήτρε οι οποίε είναι ρήτρε που περιέχουν την αμοιβαιότητα. Η κατάσταση των χωρών αυτών <clears throat> δεν πρέπει να θίξει τις κοινωνίες των χωρών αυτών που μπορούν να προσποριστούν ωφέλη από, αυτή την, ε, από αυτές τις συμφωνίες. Μέσω αυτής της ρήτρας λοιπόν μπορούμε να έχουμε ένα επικοδομητικό διάλογο για τα θέματα αυτά. Όπως είπα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να διατηρήσουμε το θέμα αυτό σε συζήτηση. Το έγγραφο το οποίο έχω παρουσιάσει θα είναι έτοιμο στις 27 του μηνός και θα έχει λοιπόν τη δυνατότητα των σύνολο των πολιτικών ομάδων να καταθέσουν τροπολογίες. Μας πιέζει το χρονοδιάγραμμα για το χρονικό σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε τη δική μας γνωμοδότηση σε άλλες επιτροπές. Θα ήθελα να διτηρήσουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα το οποίο αναφέρεται μέχρι τις 12 Ιουλίου πρόθεσμη για τις τροπολογίες και όπως έλεγε η κυρία Μουνίθ, εγώ θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη και τις θέσεις των άλλων επιτροπών. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να λάβω υπόψη τις θέσεις και τις ανησυχίες των μελών της δικής μας επιτροπής. Ευχαριστώ of July, but he said August. You have seen the... Λοιπόν, είδατε το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των τροπολογιών. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ και κλείνει η συζήτηση αυτή. Περνάμε τώρα στο θέμα του νέου πρέσβη μας στην Αλγερία, ο κύριος Σκολίλα. Έχετε το λόγο κύριε Σκολίλα.